Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε. Είναι τιμή και χαρά μου που μπορώ να υποδεχτώ εδώ την κυρία Μαγκλέιτ, που γνωρίζουμε όλοι καλά. Είναι Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Την υποδεχόμαστε εδώ σήμερα το απόγευμα με μεγάλη χαρά. Θα μας παρουσιάσει πρώτα την ε, κατάσταση και θεώρηση του περιβάλλοντος της Ευρώπης για το 2010 και μετά θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Ελπίζω και ο καθηγητής Κούλας και ο και επίσης θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ κύριε Μαγκλέτε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα το απόγευμα για να σας παρουσιάσω την ε, τέταρτη έκθεση για την κατάσταση και θεώρηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη για το 2010. Ως ευρωβουλευτές και συνομοθέτες όσον αφορά την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, ε, έχετε διαπιστώσει πόσο σημαντικός έχει γίνει ο ρόλος σας και πόσο σημαντικός πρέπει να συνεχίσει να είναι. Σήμερα, όπως ερχόμουν στο Κοινοβούλιο, σκέφτηκα ότι μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία. Πέρα από την έκθεση αυτή καθεαυτή. Υπάρχει ο τόμος που ονομάζεται η σύνθεση, που αποτελεί όντως μια συνθετική ανάλυση που βασίζεται σε διάφορα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα στις τάσεις που υπάρχουν. Έχω εδώ κάποια αντίγραφα, αλλά και σε ψηφιακή μορφή υπάρχει στη διάθεσή σας θα φροντίσω να έχουμε και άλλα αντίτυπα. Έπειτα, υπάρχουν οι θεματικές μας αξιολογήσεις, 13 στον αριθμό, που εξετάζουν τα διάφορα θέματα σε λεπτομέρειες, την εκτίμηση, την εφαρμογή, επιτυχίες και αποτυχίες. Και, πολύ σημαντικό επίσης, έχουμε και μια αξιολόγηση 38 χωρών. Είναι μοναδική περίπτωση αυτή. Έχουμε συνεργαστεί θέλοντας να έχουμε τέτοιες ενημερωμένες εκθέσεις κάθε χρόνο, ίσως και πιο συχνά ακόμα, ώστε εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις να έχουν ε, πρόσφατες πληροφορίες στη διάθεσή τους. Πολλά δηλαδή έχετε να διαβάσετε και να μάθετε. Θα περάσω στα συμπεράσματα, αλλά Επαναλαμβάνω ότι στην αρχή θα βρείτε, τη σύνθεσή μας, θα βρείτε κάποια μηνύματα κλειδί. Θα έλεγα ότι το κύριο μήνυμα είναι ότι λειτουργεί η περιβαλλοντική πολιτική. Υπάρχει πρόοδος, αλλά πρέπει να κάνουμε και περισσότερα, γιατί μας περιμένουν πολλές προκλήσεις. Ζούμε και λειτουργούμε όλοι μέσα σε ένα πλαίσιο όπου όλο και περισσότερα στοιχεία συσσωρεύονται. Χρειάζεται λοιπόν από κοινού προσπάθεια για να θέσουμε πρώτα απ' όλα καλά σε εφαρμογή τις πολιτικές μας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή αυτή. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι έχουμε περιβαλλοντικές ε, προκλήσεις, τις οποίες δεν μπορεί ο καθένας ε, μόνος του να αντιμετωπίζει. Κατά το παρελθόν είχαμε τις ε, εκπομπές, ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί, αλλά τώρα και στις τάσεις αντιμετωπίζουμε προκλήσεις που έχουν τεράστιο εύρος, που είναι περίπλοκες και που έχουν ε, να κάνουν με συνολικά συστήματα υγείας και περιβάλλοντος. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πολιτικοί έχουν μπροστά τους νέες προκλήσεις και πρέπει να καταλάβουν καλά τις διαδικασίες γιατί αλλιώ δεν μπορούν να προσφέρουν ε, λύσεις προς όφελος όλων. Οι 13 αξιολογήσεις που έχουμε και θα τους δείτε τους τίτλους που είναι το νερό, η βιοπικιλότητα κλπ έχουν να κάνουν με τις τέσσερις ε, προτεραιότητες που είναι οι κλιματικές αλλαγές, η φύση και η βιοπικιλότητα, η φυσική πόρη και τα απόβλητα και τέλος περιβάλλον, υγεία και ποιότητα ζωής. Υπάρχουν ε, οι περιλήψεις, φαντάζομαι ότι έχετε πάρει όλοι τα έγγραφα που ετοιμάσαμε για τις τέσσερις αυτές θεματικές ενότητες. Και βλέπετε ότι Μιλάμε για την πρόοδο που έχουν πετύχει 27 χώρες για να πετύχουμε τους στόχους ε, του Κιώτο. Στη σύνθεσή μας θα δείτε στον πίνακα 1-2, στις σελίδες 18 και 19 αν δεν απατώμε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που εξηγούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει όντως πρόοδος, ότι έχουμε πετύχει κάποιους στόχους, αλλά σε άλλους στόχους δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να ε, αντιμετωπίσει και να καλύψει τους στόχους του πρωτοκόλου του Κιώτου εν ώψη του 2002 με τους στόχους που έχει βάλει για τις εκπομπές. Όμως, παρόλο που η γενική τάση είναι θετική, επιμέρους δεν είμαστε θετικοί. Στις μεταφορές, για παράδειγμα, όχι. Η Λευκή Βίβλος είναι κάτι που πρέπει όλοι να προσέξουμε όλους ιδιαίτερως. Μιλώντας χτες με την Γενική Διευθύντρια, διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να επηρεάσουμε την κατάσταση εκεί. Γενικά μιλώντα, όμω, πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, τώρα που ξεκινάει και το Κανκούν, ότι οι διεθνεί προσπάθειε που γίνουν για να μειωθούν οι εκπομπέ ε, του αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ε, αύξηση της θερμοκρασίας και να είναι αυτή κάτω από δύο βαθμούς. Όσον αφορά τώρα τη φύση και τη βιοπικιλότητα, η Ευρώπη έχει πετύχει κάποια πρόοδο, όπως γνωρίζετε όλοι. Δεν μπορέσαμε όμως να πετύχουμε τον στόχο αυτό καθεαυτό. Βέβαια η Natura 2000 καλύπτει 18% της ε, γης, οι νομοθεσίες για τον αέρα και το νερό μείωσαν ε, την πίεση στην ε, βιοπικιλότητα. Όμως πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να πετύχουμε περισσότερα. Τουλάχιστον είμαστε σε θέση να πούμε ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα γιατί δεν πετύχαμε τους στόχους μας μέχρι τώρα. Τι φταίει στη βιοπικιλότητα, για τα διάφορα είδη, για την οδηγία των οικοτόπων κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, σχετικά με τον στόχο που έχει μπει όσον αφορά για τα διάφορα είδη που αναφέρονται στην οδηγία για τους οικοτόπους, ε, δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τους φυσικούς πόρους τώρα και τα απόβλητα. Και εδώ κάνουμε κάτι, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει πρόκληση. Γιατί χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερους σπόρους και άρα χρειαζόμαστε ένα καλύτερο τρόπο για την απορρόφηση των τρων εκατομμυρίων αποβλήτων που έχουμε. Για την ποιότητα ζωή τώρα, το περιβάλλον και την υγεία. Εδώ έχουμε κάποια πρόοδο όσον αφορά τα οξύδια του αζότου, τον μόλιβδο, το μονοξύδια του αζότου, το θείο. Όμως ανησυχίες για την υγεία παραμένουν. Η επεξεργασία υδάτων επίσης είναι κάτι που παραμένει. Έχουμε εντοπίσει τις πηγές μόλυνσης των υδάτων με χημικά και άλλες ουσίες που έχουμε καταφέρει να απαγορευτούν τελευταία. Προχωράμε στο τρίτο σημείο που έχει να κάνει με την αξιολόγηση των χωρών. Εδώ υπάρχουν κάποιες απαντήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο περιβάλλον και την υγεία. Ξέρουμε πώς να ανταποκριθούμε, ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε. Εκεί όπου δεν υπάρχει πρόοδος, πρέπει να φροντίσουμε για καλύτερη εφαρμογή ή να αναπτύξουμε νέους κανόνες. Και ακριβώς εδώ είναι που υπάρχουν και οι απαντήσεις όσον αφορά τα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις χώρες. Είναι περίπλοκα εδώ τα θέματα και όπου υπάρχουν επιβαλλοντικέ πολιτικές πάνε καλά. Αλλά πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως. Πράγμα το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο και δεν φαίνεται και πάντα από την αξιολόγηση που γίνεται στις χώρες για το πόσο καλά εφαρμόζεται η πολιτική μας. Εξαρτάται από τις ε, τοπικές συνθήκες. Είσαστε ευρωβουλευτές από ολόκληρη την Ευρώπη και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Ελπίζω η εξολόγηση που έχουμε κάνει εμείς να μπορέσει να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μας. Η έκθεσή μας λοιπόν για το 2010 χρησιμοποιεί την εξολόγηση αυτή των χωρών ώστε να συγκεντρώσουμε στοιχεία από τις διάφορες χώρες σε μια κεντρική δομή και να μπορέσουμε έτσι να μάθουμε ένας από τον άλλον. Είναι ένας τεράστιος πλούτος πληροφοριών. Από εκεί φαίνεται τι λειτουργεί καλά, τι δεν λειτουργεί καλά, τι δεν λειτουργεί καλά σε ένα συγκεκριμένο μέρος και τι αντίκτυπο έχουν οι πολιτικές μας. Σας ανέφερα ποιες είναι οι τάσεις στο τμήμα Α, αλλά εδώ υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Δείχνει ότι το περιβάλλον στην Ευρώπη, όπως συμβαίνει και με τις κοινωνίες και με την οικονομία, επηρέάζεται από πολλούς παράγοντες. Γι' αυτό και υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Πρέπει συνεπώς να επιταχύνουμε το feedback, δηλαδή να έχουμε μια ανάδραση, να ξέρουμε τι συμβαίνει για να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση σε διάφορους τομείς. Τώρα η διαχείριση των κινδύνων που υπάρχει τώρα που είμαστε σε μια περίοδο τεράστιων αλλαγών είναι μια παραπάνω πρόκληση. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα κλειδί και εδώ. Να βελτιώσουμε τις προβλέψεις μας για τις μελλοντικές ε, αλλαγές. Να μην αναλύουμε βάση του τι συμβαίνει σήμερα, αλλά να προκαταλάβουμε το μέλλον. Καλό σχεδιασμό επίσης. Θέλω να διασφαλίσουμε ότι όταν έχουμε μπροστά μας περιβαλλοντικές πολιτικές να μπορούμε να συνδέσουμε τις μεγάλες τάσει μεταξύ τους και να φροντίσουμε άλλες πολιτικές που παρεμβαίνουν, εμπόριο για παράδειγμα, εξωτερική βοήθεια κτλ. να μπορούν να παίξουν και εκείνε κάποιο ρόλο έτσι ώστε να προσφέρουμε περισσότερα για το περιβάλλον αντί να έχουν αρνητικέ συνέπειε. Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των προκλήσεων, είναι σαφέ ότι χρειαζόμαστε και περίπλοκες ε, λύσει στι πολιτικέ μας, όπου να συμμετέχουν όλοι οι τομείς. Διαβάζοντας τη σύνθεση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιος ε, σκοπός. Περισσότερες πληροφορίες πρώτα απ' όλα χρειάζονται για τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Ποιο είναι το κεφάλαιο που διαθέτουμε, ε, καταστρέφεται αυτό ή πώς προστατεύεται ανάλογα με τις αλλαγές του κλίματος. Ρόλος μας δεν είναι να κάνουμε προβλέψεις ε, για καταστροφές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μέλλον του περιβάλλοντος να συνδέεται με το μέλλον της γεωργικής πολιτικής, ελευτικής πολιτικής κλπ. Δύο σημεία θα αναφέρω τέλος. Το ένα έχει να κάνει με την αβαχίδα μας, που είναι η αυτάρκειά μας. Εδώ χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαχειριστούμε καλά τα αποθέματα που διαθέτουμε, να φροντίσουμε να τα διατηρήσουμε και από την άλλη μεριά ε, να δούμε και την κοινωνία. Η αυτάρκεια, ευρέως ε, ορισμένη, σημαίνει ότι τα οικοσυστήματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τους πόρους που χρειαζόμαστε. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, να έχουμε μια βιώσιμη κατάσταση στο μέλλον, είναι να είμαστε αυτάρκεις. Σε ένα βαθμό. Υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ εδώ και είναι το κατά πόσο τελικά που χρησιμοποιούμε, να δούμε από πού έρχονται. Τι διαπιστώνουμε, ότι ένα από τα μηνύματα κλειδί είναι ότι είμαστε βαθιά εξαρτημένοι αντί να είμαστε αυτάρκεις. Εξαρτόμαστε από τα αγαθά τα οποία ε, φέρνουμε από αλλού. Είτε πρόκειται για τα καύσιμα, πρέπει να προσπαθήσουμε ζήτηση και προσφορά να βρίσκονται σε κάποια ισορροπία. Και αυτό θα μας βοηθήσει να περάσουμε στην πράσινη οικονομία. Η πράσινη οικονομία έχει πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς. Και ο κίνδυνος είναι βγαίνοντα από την οικονομική ύφεση να συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε και πριν. Δεν θα έπρεπε όμως. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ε, κατευθυντήριες γραμμές προς μια νέα κατεύθυνση, για μια πραγματική ε, πράσινη οικονομία. Χρειάζεται λοιπόν ε, να έχουμε πάρκια πόρων για να πετύχουμε αυτή την πράσινη οικονομία. Πλέον έχουμε και την... το θέμα της συνοχής των πολιτικών μας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντι στις προσπάθειές μας για το περιβάλλον και όχι να το καταστρέφουμε απαλού. Χρειάζεται συνεκτική πολιτική λοιπόν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά μιλώντας υπάρχει συνοχή. Βέβαια στη θεωρία φαίνονται καλά τα πράγματα. Ήδη όμως βλέπουμε ότι διαπιστώνονται δυσκολίες και όταν εφαρμόζουμε τη θεωρία στην πράξη, πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Για παράδειγμα, το θέμα της ε, τιμολόγησης του ύδατος. Μπορεί τελικά να διαπιστώσουμε ότι η ποσότητα και η συγκέντρωση των παραγόντων που καταστρέφουν το νερό έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν ότι μέσα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πρέπει να τα έχουμε σκεφτεί καλά. Πώς βελτιώνεται η συνοχή. Όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς, έτσι και στο περιβάλλον, πρέπει να δούμε σε τι επίπεδα εφαρμόζουμε πολιτικές για το περιβάλλον. Η διαδικασία λοιπόν που ακολουθήσαμε για να αξιολογήσουμε την κατάσταση στις διάφορες χώρες έχει σαν αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και να βοηθήσουμε έτσι και εσάς να μπορέσετε να νομοθετήσετε καλύτερα. Η έκθεση σας ε, βοηθάει με την αξιολόγησή της να σχηματίσετε μια εικόνα για τα διάφορα θέματα σε διάφορες κλίμακες και να σας δώσει μια καλύτερη εικόνα του πολύπλοκου συστήματος που έχουμε με τα διάφορα επίπεδα. Και σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγέ όσον αφορά το κλίμα, ε, θέματα όπως έχουν να κάνουν με το νερό και τον αέρα, περιλαμβάνονται στους στόχους μας για το 2020. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα τους πετύχουμε αυτούς, στον κάθε στόχο ξεχωριστά, αλλά και σε συνδυασμό των στόχων αυτών. Στηρίζουμε την δουλειά της Επιτροπής για νομοθεσία όσον αφορά την αυτάρκεια πόρων. Μαζί σας θέλουμε να διερθώσουμε καλύτερα. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό ρόλο. Άρα και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα διάφορα επίπεδα ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ο καθένας έχει να παίξει το δικό του ρόλο, έτσι ώστε η χρήση πόρων από το περιβάλλον να γίνεται ε, με λογικό τρόπο και αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ την εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Πολύ σαφής και ακριβής η παρουσίασή σας και νομίζω ότι θα ακούσουμε πολλές ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ξεκινώ δίνοντας το λόγο στον ε, κύριο Γκέρμπεν Γιάν Γκερμπράντι, που είναι και το σημείο επαφή μα με τον οργανισμό και που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Μακλέιτ, για την παρουσίασή σα και για την εξαιρετική έκθεση που μα κάνατε. Δεν μιλάμε μόνο για την ε, σφιγμομέτρηση ε, της Ευρώπης και για την ε, θερμοκρασία στην Ευρώπη αλλά και για μας συγκεκριμένα γιατί νομίζω ότι σφιγμομετρώντας τις αντιδράσεις μας βλέπουμε ότι ε, είναι αποτελεσματική η πολιτική για το περιβάλλον στην Ευρώπη. Έχω κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Μιλήσατε για την εφαρμογή, για την υλοποίηση και είπατε ότι πρέπει να επιταχύνουμε την υλοποίηση. Αυτό τι σημαίνει. Ότι αφενός μεν μπορούμε κάπως να χαλαρώσουμε την νέα νομοθεσία και να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας ε, στην ε, επιβολή της νομοθεσίας και την υλοποίηση αυτών που ήδη έχουμε. Και αυτό σημαίνει παράλληλα ότι αν τα κράτη-μέλη είχαν υλοποιήσει την νομοθεσία όπως ε, υποτίθεται ότι έπρεπε να είχαν κάνει, το περιβάλλον θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε με αυτού. Δεύτερο σημείο. Είπατε ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε ένα πακέτο ε, που θα λαμβάνει υπόψη και την αποτελεσματικότητα των πόρων. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην αγορά τώρα είναι ότι οι εταιρείε προσπαθούν να ακολουθήσουν βιώσιμη ανάπτυξη λόγω οικονομικών αιτίων, όχι για κανένα άλλο φιλοσοφικό μέλημα και η σπάνιση των πόρων αλλάζει τον τρόπο παραγωγής προϊόντων και για τις εταιρείες. Νομίζετε εσείς ότι αυτή τη στιγμή οι αγορές κινούνται ταχύτερα από ότι οι κυβερνήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί. Είναι δύσκολο να προκύψουν νέε προτάσει σε μεγάλε διασκέψει των Ηνωμένων Εθνών, παραδείγματο χάρη, ενώ οι εταιρείε φαίνεται ότι κινούνται ταχύτερα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τον συναδελφό μου, τον Τζοκ Μάρτιν, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και στην παρουσίαση όλων αυτών. Θα του δώσω το λόγο λοιπόν για τις διάφορες χώρες και θα επανέλθω κι εγώ ίσως για τη γενικότερη πολιτική. Yes, with respect to the... Uh, Όσον αφορά την ερώτησή σας για την υλοποίηση αν δείτε τη συνολική αξιολόγηση των 27 κρατών μελών και των 5 χωρών ΕΖΕΣ, συν των 6 χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αποκομίζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Παραδείγματο χάρη, είναι ενδιαφέρον να δούμε τη σχέση μεταξύ της πρόοδου υλοποίησης και του μεγέθους της χώρας. Συχνά διαπιστώνουμε ότι οι μικρότερες χώρες με απλούστερους ε, μηχανισμούς διακυβέρνησης ε, προχωρούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από ότι μεγαλύτερες χώρες με ομοσπονδιακή δομή. Η εικόνα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μας δείχνει ότι με τους σωστούς όρους, τις σωστές προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών προϋποθέσεων μπορεί να σημειωθεί σημαντική πρόοδος και αυτό αντανακλάται και στις δράσεις ε, που αναλαμβάνουν και στις εκθέσεις πρόοδου για τις δράσεις αυτές. Πολύ σημαντικό είναι να διδασκόμεθα ημένα ε, από τους ΔΕ και να μπορούμε να προωθήσουμε προγράμματα αδελφοποίησης και να υποφελούμεθα από τις βέλτιστες πρακτικές. Σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών, Γνωρίζουμε ότι σε εποχές οικονομικής ύφεσης τίνει να φύγεται το περιβάλλον λόγω δημοσιονομικών μειώσεων σε αυτό το τομέα σε σχέση με άλλους τομείς. Όμως είναι επίσης σαφές ότι ε, υπάρχει και ολοκλήρωση των πολιτικών που είναι διαφορετική στο βορρά της Ευρώπης από ό,τι στο νότο της Ευρώπης. Και όταν βλέπετε τέτοιες πολιτικές ολοκλήρωσης, αυτό αντανακλάται στη διαδικασία επιτάχυνσης. Για την ερώτηση λοιπόν σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίηση. παίζει σημαντικό ρόλο η προοπτική της ε, ενοποίησης και ολοκλήρωσης. Βλέποντα τι εκθέσει για τις μεμονωμένε χώρες, δεν βλέπουμε καθόλου ότι θα ήταν κάτι το ευκταίο το να έχουμε χαλάρωση των πολιτικών για τον περιβάλλον σε οποιαδήποτε χώρα εξετάσαμε στην αναλυσή μας. Αντιθέτω, βλέπουμε ότι αυτό που θα ήταν προτιμότερο είναι μεγαλύτερη σαφήνεια για το τι απαιτείται στην υλοποίηση και σε μεγάλο βαθμό απλούστευση απλοποίηση αυτών τα οποία απαιτούνται. σε πολλούς τομείς όταν ε, εξετάζουμε τις περιβαλλοντικές πολιτικές συγκρίνοντάς τις με τις διάφορες τομεακές ε, ε, πολιτικές βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλαπλά αιτήματα σε θέματα περιβάλλοντος και δεν γνωρίζουν οι αρμόδιοι φορείς πώς να ερμηνεύσουν αυτά τα αιτήματα και δεν είναι σαφές πώς θα τα υλοποιήσουν κατά τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Άρα υπάρχει μια σχέση μεταξύ σαφήνειας και απλούστευσης που θα μπορούσε να είναι ισόφελος της διαδικασίας επιτάχυνσης. Η ε, κυρία Μακλέη. Για τη συνολική πολιτική για το περιβάλλον θα δείτε και στην έκθεση πολλές απαντήσεις από αυτού, αλλά θα προσπαθήσω να το συνοψίσω. Ο λόγος για τον οποίο οι αγορές αυτές καθεαυτές προσπαθούν να είναι αποδοτικές και αυτό το έχουν κάνει επίκεντρο της πολιτικής τους. Βλέπουμε ότι είναι σημαντικό ε, να φροντίσουν να έχουν χαμηλό κόστος και για τα υλικά τους και για τον εφοδιασμό τους και αντιλαμβάνονται οι εταιρείε που ασχολούνται με αυτά τα θέματα ότι η Ευρώπη έχει σπάνιδα πόρων και επομένως αυτή η πόρη είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό προσπαθούν οι εταιρείε να γίνουν αποδοτικέ ε, σε σχέση με του πόρου που χρησιμοποιούν. Και κάνοντα μια προβολή και στο μέλλον, βλέπουμε ότι προχωρούμε με το σωστό τρόπο. Βλέπουμε αύξηση τη αποτελεσματικότητα, μείωση τη ρήπανση ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα σε διάφορε περιοχέ. Και βλέπουμε ότι αναπτύσσεται ο συνολικό όγκο τη οικονομία παράλληλα. Και ένα δείκτη που είναι ενδιαφέρον ε, είναι σε σχέση με την καινοτομία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στην Ευρώπη, αλλά αν δούμε την κατάσταση στην Κίνα, βλέπουμε ότι είναι τεράστια η αύξηση στην Κίνα. Και για μας είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα, διότι παρά τις πολλές μας προσπάθειες, ε, δέχεται να μπούμε σε ένα διάλογο για το ποιος κάνει τι στη μεταφορά τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα που αξίζει να προσέξουμε. Κάποιοι τομεί, κάποιοι κλάδοι ε, ε, είναι προηγμένοι, τώρα δεν ξέρω αν οι κοινωνίε θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι εν μέρη μια απάντηση για θέματα πολιτικής και οράματος. Ευχαριστώ πολύ. Chris Davis. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κυρία Μαγκλέιντ. Χαίρομαι ε, που σας ακούω και χαίρομαι που μπορώ να κάνω και τις ερωτήσεις μου για, τις, για τα θέματα κλιματικών αλλαγών. Καταρχάς, η έκθεση μας λέει ότι είμαστε στην πορεία μέχρι το 2020 να περιορίσουμε τις εκπομπές μας. Ταυτόχρονα όμως λέει ότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν τις εκπομπές ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν τα θέματα εξαγωγών των εκπομπών. Όμως, αν κατάλαβα καλά, η καθαρή μας συνεισφορά στην, ε, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι μηδενικές, είναι μηδενική. Και μηδενική θα είναι και η συνδρομή μας, η συνεισφορά μας μέχρι το 2020. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό, διότι έχουμε εξάγει ε, τις εκπομπές μας αλλού. Επίσης, λέτε στην έκθεση ότι το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ε, θέλει περισσότερες ε, μειώσεις στις εκπομπές από αυτές που πρόβλεψε το Κιώτο. Και διαρωτώ με, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε και άλλες δυνατότητες, τα SFC ας πούμε, οι χλωροφθοροϊδρογονάνθρακες ή θα πρέπει να δούμε και άλλα θέματα αντα... αλλαγής ε, με άλλες εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή όσον αφορά επίσης και την ενεργειακή πολιτική. Τώρα, το επίπεδο της θάλασσας, τρία χιλιοστά το χρόνο ανεβαίνει ε, το επίπεδο της ε, θάλασσας. Όντως, ο Ρότσορ Χέλμεν, ένας από τους πιο σημαντικούς ε, σκεπτικιστές για την αλλαγή του κλίματος, λέει ότι πήγα σε πάρα πολλά μέρη, αλλά δεν είδα ποτέ να ανεβαίνει η θάλασσα. Ε, βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντως και εγώ δεν βλέπω να έχει ανέλεύει η θάλασσα σε ορισμένα σημεία, αλλά τέλος πάντων έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει και η άμμος και τα λοιπά. Τώρα. Μέσα σε ένα αιώνα, πώς θα φτάσουμε στο 1-2 μέτρα. Επίσης το θέμα της εφαρμογής, ότι τα κράτη-μέλη θα επωφεληθούν από μια ε, μεγαλύτερη διαφάνεια. Διερωτώ με, έχετε κάνει μια, καμία σύσταση στην, στην Επιτροπή όσον αφορά την, ε, για την εφαρμογή της ε, πολιτικής ή της εκπόνησης πολιτικής, θα πρέπει οι, οι οδηγίες να δίδονται εκ των προτέρων. Αυτό θα βοηθούσε περισσότερο. Και θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε με απλά λόγια τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Διότι φαίνεται ότι ό,τι συζητάμε εδώ δεν εφαρμόζεται σωστά από τις ε, ε, από τους αξιωματούχους, αν θέλετε, των κρατών μελών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαγκλέιντ και εσάς προσωπικά, αλλά και όλη το προσωπικό το οποίο είναι πλάκι στην, ε, στην ε, σύνταξη της έκθεσης αυτής. Δεν το έχω, δεν τη διάβασα, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι τόσο καλή αυτή η έκθεση όσο και η προηγούμενη. Μπορώ να σας πω, από προσωπική μου πείρα, ότι η Πρόκειται για μία από τις εκθέσεις που την θεωρούμε σημείο αναφοράς και στην Επιτροπή μας και στις διαπραγματεύσεις. Στο γραφείο μου ε, το χρησιμοποιεί, το βιβλίο το οποίο χρησιμοποιούμε περισσότερο για να δούμε κάτι κτλ. Πραγματικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μας έχουν βοηθήσει οι εκθέσεις σας και χαίρομαι που μπορώ να ε, περιμένω να διαβάσω την έκθεση. Θα ήθελα να κάνουμε κάποια σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εστιάζετε την προσοχή σας στην ανάγκη να, ολοκληρώσει, να ενταχθεί η περιβαλλοντική πολιτική και σε άλλες πολιτικές. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά τις επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια και στην Επιτροπή μας, αλλά και στο Κοινοβούλιο με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και με τις πολιτικές μεταφορών που αναθεωρούνται. Ε, επομένως, είναι πολύ σημαντικό η περιβαλλοντική πτυχή να μην ενταχθεί μόνο στην πολιτική περιβάλλοντος, αλλά και σε άλλες πολιτικές. Λοιπόν, οι ερωτήσει μου δεν αφορούν την έκθεση, δεν την έχω διαβάσει, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο, πόσο μεγάλη έμφαση δώσατε στη σχέση ανάμεσα στην οικονομία, στην οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον και την πολιτική περιβάλλοντος. Γιατί όπως ξέρετε ίσως πάρα πολύ καλά, τα θέματα αυτά, τα οποία συζητάμε πολύ αυτούς τους τελευταίους μήνες, το συζητήσαμε για την βιοπικιλότητα, αλλά και για το κατά πόσον θα πρέπει να ανεβάσουμε, αν θέλετε, το επίπεδο ελέγχου μας ε, στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών. Ε, όντως θεωρώ ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο φιλοδοξιών μας, όχι μόνο για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και γιατί με τον τρόπο αυτό θα αυξήσουμε και την ανταγωνιστικότητά μας. Λοιπόν, μήπως θα μπορούσατε να σχολιάσετε τα θέματα αυτά. Δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία πώς συνδέονται μεταξύ τους και τι γίνεται με τη σχέση ανάμεσα στο κόστος για την, κοινωνία σχετικά με την προσαρμογή και πώς μπορούμε να συγκρίσουμε αυτό το κόστος με την πρόληψη. Ευχαριστώ. Ο Κάρλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και κάνατε την παρουσίασή σας. Έριξα μια γρήγορη ματιά στην έκθεση τώρα. Θα ήθελα να μιλήσω για άλλα θέματα εκτό τη κλιματική αλλαγή καταρχήν, για να μην τα ξεχάσουμε. Τα χημικά καταρχήν. Έχουμε δει διάφορε τάσει για τι χημικέ ουσίε τα τελευταία χρόνια και για τα CMR και για τα τοξικά. Βλέπουμε ότι ε, αυξάνονται και οι όξινε ουσίε. Και είπατε ότι ίσως αυτά αποσυνδεθούν από την ανάπτυξη. Τι νέου είδους ε, νομοθεσία για τις χημικές ουσίες χρειαζόμαστε για να τα αποσυνδέσουμε. Με τις υψηλότερες, με τις καλύτερες γνώσεις που έχουμε ε, για, τις, ε, για τους ορμονικούς διαταρακτές υπάρχει ένα θέμα που εδώ συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Τι θα μπορούσαμε κατά τη γνώμη σας να κάνουμε που δεν έχουμε κάνει. Για την βιοπικιλότητα Όντως έχουμε νέες δεσμεύσει και τις στηρούμε, αλλά θέματα όπως ε, η χρήση γης, ε, τα πτηνά είναι διάφορα θέματα πολύ ενδιαφέροντα που κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, γιατί η τρέχουσα νομοθεσία μάλλον δεν αρκεί. Και το μεγάλο ερώτημα τελικά για την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι το πραγματικό θέμα είναι αυτό ακριβώς η αποδέσμευση. Κάπου στην αρχή της έκθεσης υπάρχει ένας πίνακας με ένα κύκλο που δείχνει τα ποσοστά εκπομπών στους διάφορους τομείς και τις μέχρι τώρα μειώσεις. Ψητικές ε, χημικές ενώσεις και απόβλητα είναι τομείς στους οποίους είμαστε επιτυχημένοι. Τώρα όμως αποτελούν πολύ μικρό τμήμα των εκπομπών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεταφορές που αυξάνονται και η παραγωγή ενέργειας και ακόμη και αν ε, αλλάξουμε ε, την πηγή για την παραγωγή ενέργειας ε, θα συνεχίσουμε να ε, έχουμε δυσκολία μείωση των εκπομπών και υπάρχουν ορισμένα θέματα που θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την αύξησή τους. Πιο δύσκολο από άλλα. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας ε, κάνετε μια παρουσία στο μέλλον ή μια έκθεση για τις συστημικές σχέσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον τομέα έρευνα στο να δούμε εκπομπέ σε συσχετισμό με το χρόνο εργασίας. Μια μελέτη δείχνει ότι αν οι Ευρωπαίοι δούλευαν τις ίδιες ώρες με τους Αμερικανούς θα αυξάνονταν οι εκπομπέ μας κατά 20%. Δεν είναι περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά βλέπουμε ότι έχει επίπτωση επί του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Είναι σημαντικό θέμα αλλά δεν έχει ακόμη αρχίσει να χρησιμοποιείται στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Σε αυτό το τομέα λοιπόν θα με ενδιαφέρει να ακούσω τις δράσεις σας. Στο κεφάλαιο που μιλάει για την αποτελεσματικότητα των πόρων λέτε ότι υπάρχει πρόοδος αλλά δεν έχουμε επιτύχει ακόμη αυτό που θέλουμε και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την κλιματική αλλαγή. Κυρία Μαγκλέη, θέλετε να απαντήσετε στις πρώτες ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε μετά με τρεις νέες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Δύσκολες οι ερωτήσεις και δεν ξέρω κατά πόσο έχω απάντηση. Φυσικά, για αυτήν την καθαρή προσφορά της ε, Ευρώπης θέλουμε φυσικά να δούμε πώς θα το υπολογίσουμε. Και θα έπρεπε ήδη να το κάνουμε. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά σήμερα δεν είμαι σε θέση να σας πω ότι συνολικά είναι μηδενικό το ίχνος. Πάντως υπάρχουν ροές για διάφορα προϊόντα. Αν μας, μας ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο, μπορούμε κατά προσέγγιση να σας δώσουμε μια απάντηση για τον άθρακα και να έχετε έτσι κάποια νούμερα. όσον αφορά την ε, άνοδο του επίπεδου της θάλασσας. Έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία των ε, πόρων και με την ε, Eurostat και με τον ΩΣΑ δουλεύουμε σε αυτό. Πάντως συγκεκριμένα για την άνοδο του επίπεδου της θάλασσας. Ναι. Βλέπουμε δείγματα ε, που περνάει το αλατισμένο νερό. Δεν έχει σημασία που ακριβώς ε, βρίσκεσαι στην ε, Ευρώπη. Εντάξει, προς την Σκοτία ανεβαίνει, τώρα δεν ξέρω εσείς που ακριβώς ζείτε. Αλλά μπορώ να σας δείξω σημεία που ήδη βλέπουμε στις ακτές μετά από δύσκολες καιρικές συνθήκες να υπάρχει τέτοια πρόοδος του θαλάσσιου νερού. Είναι λοιπόν ζητήματα με τα οποία οι μηχανικοί πρέπει να ασχοληθούν. Με το πρόγραμμα προσαρμογής μας προσπαθούμε να κάνουμε μια καταγραφή. Ελέγχουμε λοιπόν το επίπεδο της θάλασσας. Γιατί άνοδος παρατηρείται σε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς παρατηρούμε γύρω από τα λιμάνια κυρίως της Ευρώπης τι γίνεται και εκεί έχουμε στοιχεία που μας βοηθούν να κάνουμε προβλέψεις. Όλα εξαρτώνται όμως από το πόσο καλή δουλειά θα κάνουμε για να αποφύγουμε τα αέρια του θερμοκηπίου. Το Ροτσόκ θα μιλήσει περισσότερο για την εφαρμογή. Πάντως, μια που βρίσκομαι εδώ και συνεργάζομαι μαζί σας και με τους συζητητές σας. Πολλές φορές ακούμε πώς ε, θα μετρήσετε την πρόοδο από τη στιγμή που θα υπάρξει η νομοθεσία. Ε, λοιπόν, εμείς ε, σημειώνουμε όλους τους δείκτες, έχουμε πολλούς δείκτες που μας βοηθούν. Και τι βλέπουμε βλέπουμε ότι έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία και πληροφορίες για τους δείκτες που αρχικά θέλαμε, αλλά που δεν είναι αρκετοί για να απαντηθούν όλα τα δικά σας ερωτήματα. Καλό λοιπόν είναι να ξέρουμε συγκεκριμένα τι θέλουμε να μετρήσουμε. Προτείναμε και θέλουμε να μας στηρίξετε κι εσείς να βρούμε ένα σφαιρικότερο σύστημα υπολογισμού ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε και για το μέγεθος και για την ποιότητα της γης, του νερού, της βιοπικιλότητας. Και έτσι να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις επιπτώσεις πάνω σε αυτούς τους πόρους, τη γη, το νερό κλπ. Ελπίζω να τα καταφέρουμε αν βασιστούμε στην στατιστική προσέγγιση του ΟΗΕ. Όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά χρειαζόμαστε πολιτική στήριξη. Γιατί είπαμε, ότι μια μεριά έχουμε τη στατιστική και από την άλλη μεριά έχουμε το περιβάλλον. Πάντως μπορεί κανείς να ζητήσει πράγματα με την νομοθεσία που να βοηθήσουν να δούμε πιο ξεκάθαρα την κατάσταση. Αλλά θα δώσω σε λίγο το λόγο στο συνάδελφο να σας εξηγήσει περισσότερο. Για την οικονομία τώρα και την ανταγωνιστικότητα. Όπως γνωρίζετε, συζητάμε για ένα διαφορετικό ΑΕΠ και θέλουμε να συμπεριλάβουμε και άλλους δείκτες στο ΕΠ. Και ελπίζω να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και την αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής μας πολιτικής. Γίνεται ανάλυση που δεν έχει ε, δημοσιευθεί ακόμα, περιμένουμε τα Υπουργεία, να δούμε πόσο στοιχίζει η εφαρμογή μιας νομοθεσίας. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι γίνεται μια μεγάλη επένδυση στην αρχή και μετά το πράγμα μένει στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε και περισσότερα πράγματα λοιπόν για την εφαρμογή. Δεν φτάνει η αρχική επένδυση, χρειάζεται και συνέχεια για να μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα στην ποιότητα των υδάτων τα, το νερό, έχει να κάνει φυσικά με την καλλιέργεια του εδάφους και επηρεάζεται από τη χρήση των κλπ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενδιαφέροντα στοιχεία λοιπόν για να συζητήσουμε για το αλλιώτικο ΑΕΠ ή πέρα από το ΑΕΠ, το καθάριστο εθνικό προϊόν. Άπαξ και έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο και έχουμε κάποια, κάποιες κατά ουσίες, τα χημικά, οι χημικές ουσίες περνούν στο περιβάλλον έτσι κι αλλιώς. Αλλά εντοπίζονται. Καρκινογόνες ουσίες, φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά είναι ουσίες που φτάνουν στο νερό. Το θέμα του να βάλουμε μια τιμή στο νερό θα οδηγήσει ίσως στο να χρησιμοποιεί ο κόσμος λιγότερο νερό. Και έπειτα για να αποφύγουμε αυτήν την μόλυση χρειάζεται περισσότερο νερό, ακριβώ για να διαλυθούν, να γίνει πιο μικρή η συγκέντρωση αυτών των ουσιών στο νερό. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε στόχους για συγκεκριμένες χημικές ουσίες, δεν νομίζω. Νομίζω το θέμα της πηγής των πόρων πρέπει να δούμε περισσότερο να δούμε γιατί πρώτα απ' όλα χρησιμοποιούνται κάποιες χημικές ουσίες. Και έχουμε παραδείγματα. Οι γιατροί πολλές φορές για φάρμακα κάτω του καρκίνου, για παράδειγμα, προσφέρουν αναλλακτικέ λύσεις. Και προτείνουν μορφές φαρμάκων οι οποίες καταστρέφουν λιγότερο το περιβάλλον. Ευχαρίστως πάντως να συζητήσουμε περισσότερο μαζί για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τις χημικές ουσίες που περνάνε στο περιβάλλον. Για την ε, αποσύνδεση τώρα. Αν δούμε τις μεταφορές. Όταν σχεδιάζουμε για τους σιδηροδρόμους, Αν δούμε τι θα γίνει το 2050, όπου δεν θα είναι τόσο πολύ τα ορυκτά που θα χρησιμοποιούνται για ενέργεια και οι περισσότερες μορφές μεταφορών θα είναι ηλεκτρικές ε, ή θα χρησιμοποιούν κάτι άλλο, τότε πρέπει να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των υποδομών. Έγινε και ε, στις αερομεταφορές με το μέγεθος των αεροπλάνων. Έτσι και εδώ πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιεί το χώρο στην Ευρώπη. Όταν έρχεται σιδηροδρόμος και φτιάξετε περισσότερο σιδηροδρόμους, επηρεάζεται τη βιοπικιλότητα. Χρησιμοποιείτε το χώρο, δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε μορφή έχει και τα αρνητικά της. Επηρεάζει το περιβάλλον. Όσο και αν φαίνεται πιο καθαρός ο σιδηρόδρομος σήμερα, αν το συγκρίνετε συνολικά με τις άλλες μορφές μεταφορών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται και το σιδηρόδρομο με τέτοιο τρόπο που καταστρέφει πράγματι λιγότερο το περιβάλλον συνολικά όμως. Σύντομα, κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στον συνάδελφο που έχει και αυτός να προσθέσει μερικά πράγματα. Για το σημείο σχετικά με τις χημικές ουσίες, η έκθεση που κάναμε για τα φαρμακευτικά προϊόντα και το περιβάλλον έδειξε ότι από νομοθετικής πλευράς είμαστε επιτυχείς στην διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων που δεν χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζοντας την ασφαλή τους διάθεση. Και τα περισσότερα το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος προκύπτει από το βιολογικό καθαρισμό, γιατί ακόμη και ο πιο ακριβώς βιολογικός καθαρισμός δεν μπορεί να ε, συγκρατήσει τα χημικά τα οποία καταλήγουν στις ε, υδάτινες οδούς και πρέπει να δούμε ποιος πληρώνει το κόστος των υποδομών αυτών. Σχετικά με την απλούστευση, συνεχίζοντας και από αυτό που είπε η Τζάκη για το ε, δίκτυο ε, των φορέων επαγγελματικής ε, προστασίας, πρέπει να δούμε τη σχέση μεταξύ των φορέων περιβαλλοντικής προστασίας και των τοπικών φορέων για να πληρούνται οι απαιτήσει και να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον τομέα, με τους ανθρώπους επιτόπου που δεν είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για την υλοποίηση και να μπορεί να υπάρχει σωστή επαφή. Αυτό το δίκτυο μας προσφέρει δυνατότητες ε, να κάνουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 20 χρόνια και να γίνονται καλύτερες συζητήσεις και με τα διάφορα υπουργεία στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την Judith. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαγκλέιντ που ήρθε εδώ και που ε, μας μίλησε με τόσες λεπτομέρειες. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στην έκθεση, στον οδηγό, αναφέρατε ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην διατήρηση των πόρων μας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες και πιο καινοτόμες λύσεις για τους πόρους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι εμείς αντιμετωπίζουμε την καινοτομία σαν μια τεχνική, τεχνολογική λύση σε ένα ευρύτερο πρόβλημα, στα ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα. Όπως ο συνάδελφος ε, Σλούτερ δεν είναι τεχνικά τα θέματα, είναι θέματα συμπεριφοράς, τις διαδικασίες ε, θέλουμε να αλλάξουμε. Επομένως, πιστεύετε ότι την πολιτική μας ε, καινοτομία, την πολιτική καινοτομιών θα πρέπει να την ε, προσανατολίσουμε και στις κοινωνικές πολιτικές ε, για να επηρεάσουμε και τη συμπεριφορά των καταναλωτών που είναι τόσο σημαντική για την διατήρηση και τη συντήρηση των πόρων μας γιατί μια εκστρατεία πληροφόρησης απλά δεν, δεν βοηθάει. Θέλουμε να προσελκύσουμε ε, με κάποιο τρόπο την προσοχή των ε, πολιτών, να τροποποιήσουμε την ε, συμπεριφορά των καταναλωτών. Ποιες είναι οι λύσεις σε αυτό, ο Κρήτον. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίζω την κυρία Μαγκλέιντε. Θα ήθελα να ρωτήσω πολλές να κάνω πολλές ερωτήσεις για τα δάση, αλλά ξέρετε... Αλλά αύριο έχουμε την ακρόαση για τα δάση και η κυρία Μαγκλέιντ θα μιλήσει. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος για την αναμεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, θα αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για πολλές αλλαγές που θα αποτελέσουν ούτως ή άλλως και θέμα συζητήσεων. Θα πρέπει εκτός από την αρχή ο, πληρώ, ο ρηπαίνων πληρώνει και ο επωφελούμενος να πληρώνει, να πληρώνει ταυτόχρονα. Για τις ορισμένες ευρωπαϊκές αστικές περιοχές θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση για τι εκεί είναι το πρόβλημα και όχι στις περιοχές της υπαίθρου. Χρειαζόμαστε κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία. Τα έχουμε και αν όχι, τι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μαγκλέιντε. Σας ευχαριστώ για αυτή την τόση παρουσία, για αυτή την παρουσίαση, την οποία όμως έχασα γιατί είχα καθυστέρησα. Αλλά πρέπει να ήταν εξαιρετική παρουσίασή σας ως συνήθως για την ε, κατάσταση του περιβάλλοντος. Έχω κάποιες ιδέες να, να τις μοιραστώ μαζί σας, δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Πραγματική ε, ε, δουλειά αυτή. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη τώρα και μας δίνεται και κάποια στοιχεία για τα κρίσιμα θέματα για το μέλλον. Βέβαια πρέπει να, να συνδέσουμε τα θέματα αυτά με τις πολιτικές που πρόκειται να εφαρμόσουμε στην Ευρώπη. Και υπάρχουν πολλές πολιτικές και νομίζω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα μας βοηθήσει για την ε, εκπόνηση αυτών των πολιτικών, για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ε, προφανώς δεν θα ζητήσουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ε, συμβουλές για το τι θα γίνει για τα εισοδήματα πούμε, των πολιτών. Όμως για τη βιωσιμότητα των, ε, της, διατροφ, της διατροφικής προμήθειας ε, αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορεί να μας βοηθήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ή για την βιωσιμότητα της διατροφικής ασφάλειας. Εκεί όντως νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει το ίδιο και για τις πολιτικές συνοχής και οι πολιτικές συνοχές, συνοχής της Ευρώπης θα αξιολογηθούν και ενδεχόμενα να αλλάξουν κιόλα. Αλλά το πρόβλημα είναι τι εννοούμε με περιβαλλοντική ε, ανάπτυξη και με την ένταξη της, ε, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής πτυχής στην ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή τι σημαίνει εάν η ένταξη του περιβάλλοντος στις πολιτικές συνοχής. Εκεί η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος θα είναι σημαντική. Επίσης για την πολιτική έρευνα, συζητάμε πολλά για την πολιτική έρευνα, όμως ένα από τα βασικά θέματα που ανα, που αναφέρεται και εδώ, είναι η αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αλλά τι σημαίνει η αποτελεσματική χρήση των πόρων και πώς θα μπορούσε να τον ρόλο της Ευρώπης εδώ. Υπάρχουν πιο, ε, ε, πιο εστιασμένα σημεία που θα, η συνεισφορά σας θα ήταν πολύ χρήσιμη. Επίσης, ένας άλλος τομέας που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι η, η ακρίβεια και η σαφήνεια της, ε, της Κομισιόν. Αύριο θα υπάρχει μία ανακοίνωση για τις πρώτες ύλε, για το πώς θα έρθουν οι πρώτες ύλε στην Ευρώπη. Είναι γεωπολιτική έκθεση. Επίσης ε, θα υπάρχει και μια ανακοίνωση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων το Δεκέμβρη. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ε, μια σχέση ανάμεσα στην ορθολογική χρήση της έρευνας και στις, πολιτικές, και στην, ε, και στις πρώτες ύλες. Το Σεπτέμβριο επίσης η Κομισιόν θα κάνει μια ανακοίνωση για την ανάπτυξη που θα στηρίζεται στα θέματα βιομάζας κτλ. Τι σημαίνει αποτελεσματική χρήση της βιομάζας, γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για την ιατρική, για τροφή, για τρόφιμα, για ξυλία, για ενέργεια. Επί του παρόντος όμως έχουμε μόνο σαφείς στόχους για την ενέργεια, που είναι ο πλέον αναποτελεσματικός τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα. Επομένως, εάν δούμε τη συνολική παραγωγή της χρήσης της βιομάζας, εδώ εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε τις πρώτες ύλες την έρευνα και, την, και τα βιοπροϊόντα προϊόντα, αν θέλετε. Επίσης το, το σφαιρικό παγκόσμιο κεφάλαιο με ικανοποιεί, με, με, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να ξέρω είναι ποιες είναι οι συνέπειες των κοινοτικών πολιτικών σε τρίτες χώρες. Αναφέρω την συντομία. Αν όμως θέλουμε να συζητήσουμε για τις αλλαγές ε, της πολιτικής, ε, ε, ε όταν βλέπουμε, εξετάζουμε τον, ε, την, ε, τον αντίκτυπο των πολιτικών μας, τον, τον εξετάζουμε μόνο στην Ευρώπη. Ας δούμε όμως τι γίνεται και έξω από την Ευρώπη για την, την βιοπικιλότητα, για τις εκπομπές. Ε, θα μπορούσατε και εσείς να βοηθήσετε εμάς τους πολιτικούς να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των πολιτικών μας εκτός της ε, ευρωπαϊκής επικράτησης. Γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε, ε, ξεχνάμε αυτή την πτυχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Μαγκλέιντε, να απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις και μετά θα συνεχίσουμε. Και μετά θα μιλήσει και ο κύριος Σκουλός. Κυρία Μαγκλέιντ. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις ε, και προσφέρονται για μεγάλη συζήτηση. Αυτό που βλέπουμε στη συζήτηση για την αλλαγή συμπεριφορά είναι βεβαίω ένα συγκεκριμένο σημείο και έχει σχέση και με την ερώτηση του Κάρλ για το χρόνο εργασία και το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατανόηση των βασικών μηνυμάτων τη έκθεσή μα. Έχουμε παράλληλα με τα μεγάλα επίβολα προγράμματά μα ε, και ένα άλλο τομέα που δεν θα τον έλεγα low-tech, χαμηλή τεχνολογία, αλλά τρόπο με τον οποίο μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στου πολίτε, να δούμε πώ μπορούμε να οργανώσουμε την καθημερινή δουλειά μας, τον χρόνο εργασίας μας κλπ. Οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κατανοήσει το θέμα της κινητικότητας, παραδείγματος χάρη. Και έχουμε δουλέψει του θέματος και δείχνει η εργασία μας ότι οι πολίτες είναι πρόθυμοι να εξετάσουν αλλαγές στην κινητικότητά τους τοπικά, αλλά ε, δεν είναι τόσο ανοιχτή στο να κάνουν συμβιβασμού ε, σε διακοπέ, παραδείγματο, στην κινητικότητά του όσον αφορά μεγαλύτερε αποστάσει. Είναι θέματα λοιπόν που πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε. Σε όλε τι συζητήσει που κάνουμε στου διάφορου τομεί, υπάρχει μια αντίδραση τοπική και άμεση που πρέπει να την προωθήσουμε στι τοπικέ αυτοδιοικήσει και στου πολίτε του ίδιου, ε, γιατί νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε πολύ περισσότερα. Και σε σχέση με αυτό που έλεγε ο προηγουμένω ε, για το κόστο αδράνειας είναι πολύ ψηλό το κόστο του να μην κάνουμε τίποτα. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν προωθούσε την αντίδρασή τη ε, η Δανία για τα θέματα τη κλιματικής αλλαγής για να απαλλαγούν από τα ορυκτά καύσιμα. Ξεκινώντας το 2050 και προς τα πίσω, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρά πολιτικών που αλληλοσυνδέονται χωρίς να δημιουργείται κοινωνική αστάθεια, δηλαδή μικρά βήματα σε συνδυασμό με μεγάλα βήματα και όχι τεράστιες αλλαγές που αποσταθεροποιούν το σύστημα. Ακούγοντα τι συζητήσει για τι μεταφορέ και για την ενέργεια, υπάρχει ένα κίνδυνο ε, ότι ο συνδυασμό τιμών θα μπορούσε να μα οδηγήσει πολύ γρήγορα σε μια ε, αλλαγή πηγή καυσίμων που θα ήταν ευνίδια πολύ πιο ευνίδια από ότι αν είχαμε συνεχώ μικρέ αλλαγέ σε μια δεκαετή, δεκαπενταετή, εικοσαετή περίοδο. Και αυτό είναι σημαντικό να το δούμε και για τις αλλαγές συμπεριφοράς και για τις συστημικές αλλαγές που πρέπει να βάλουμε σε ένα κατάλογο και να προωθούμε σιγά σιγά για το τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση και με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και με την ασφάλεια των τροφίμων και τη χρήση γης κλπ. Βλέπουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν ευκαιρίες. Με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι η ασφάλεια της παραγωγής τροφίμων. Και αν δούμε το ίχνος ε, και το θέμα των εκπομπών ε, διοξιδίου, μεγάλο μέρος αυτών οφείλονται στον τρόπο παραγωγής και εισαγωγής ε, ειδών διατροφής. Αν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και πιο παραγωγικά τα εδάφη και να μην κάνουμε τόσο εκτεταμένη χρήση γης ε, που μας ενδιαφέρει και για θέματα βιοπικιλότητας, βλέπουμε τις σχέσεις που υπάρχουν και με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αφενός μεν πρέπει να έχουμε ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες, που αποτελείται όμως από διαφορετικό συνδυασμό τιμών αγοράς, δηλαδή αγρότες που παράγουν τα τρόφιμά τους κοντά στις πόλεις, και αν το ε, συνδέσουμε με αγρότες που βρίσκονται στην περιφέρεια, με μικρότερη πρόσβαση στην αγορά, που όμως ε, παρέχουν ένα δημόσιο αγαθό διότι διαχειρίζονται τη γη και είναι ε, πολύ θεωρητικό το έργο τους για θέματα βιοπικιλότητας κλπ. Αν με ρωτήσετε το πού θέλουμε να παρέμβουμε σε σχέση με το δίκαιο εισόδημα και το περιβάλλον, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το να δώσουμε ποσοτικά δεδομένα που θα αποδεικνύουν πού μπορούμε ε, να προωθήσουμε το σωστό προγραμματισμό για να χρησιμοποιήσουμε τα εδάφη που έχουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις ικανότητες που έχουμε για τη βιοπικιλότητα. Και εδώ είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε συνεκτικά και συνδέεται και με το θέμα του ύδατος και του ποιος επωφελείται από τον πόρο αυτό. Αυτές είναι κάποιες γενικές ιδέες που έχουμε, όπως επίσης και το να ασχοληθούμε με το θέμα της βιομάζας και στον τομέα της ενέργειας, ε, γιατί θα παίξει το ρόλο της η βιομάζα, αλλά πάλι θα θεωρείται ως κάτι το οποίο καταλαμβάνει χώρο, καλύπτοντας ε, ένα χώρο και θα πρέπει να είναι ένας από τους παράγοντες επιλογής για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις κλπ. Και θα δώσω πάλι το λόγο στον Τζοκ για να μιλήσει για τους, για τους ωφελούμενους και για το ποιος πληρώνει και ποιες είναι οι οικονομικές απαντήσεις που μας ενδιαφέρουν για το μέλλον. Λίντα Μαγκάουαν. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, να δώσουμε το λόγο στον συναδελφό σας πρώτα. Για τους δικαιούχους, για τους επωφελούμενους, ε, θα είναι σύντομος ε, στα σχολιά του συνάδελφος. Κάνοντας τους υπολογισμούς μας, εξετάσαμε δύο σχετικά θέματα. Πρώτον, για την επίπτωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω, όπου εξετάζουμε ε, την ε, γη η οποία έχει αφιερωθεί στα 144 περισσότερο καλλιεργούμενα γεωργικά προϊόντα Μπορούμε λοιπόν να δούμε τις εμπορικές ροές από πλευράς χρήσης γης και βλέπουμε ότι η καθαρή εξάρτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,6 εκατομμύρια εκτάρια ανά έτος. Αυτό είναι μια υπολογιστική τακτική. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτά τα θέματα και να κάνουμε πιο πολύπλοκους υπολογισμούς αν θέλετε. Το θέμα για το κατά πόσο μπορούμε, μπορεί αυτή η περιφέρεια να συνεχίσει να βασίζεται αξιόπιστα στο ίχνος του άνθρακα που έχουμε είναι μια μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όταν κάνουμε το διάλογο για τα θέματα αυτά για να έχουμε δική μας μέθοδο υπολογισμού για το ίχνος ε, των ε, ειδών διατροφής. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε τον πρώτο πίνακα ε, για τα, κράτη -μέλη της 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εισρωές και εκροές για τις εκπομπές διοξίδου του άνθρακος και για διάφορους πόρους και αυτό ανοίγει ενδιαφέρουσες δυνατότητες για το ποιος ωφελείται από τη χρήση της φύσης. Διότι στο ΑΕΠ οι πρωτογενείς τομείς, γεωργία, λία, δασοκομεία, αποτελούν το 3% του συνόλου για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν υπολογίσουμε και το ποιος χρησιμοποιεί το προϊόν της δασοκομείας, της αλίας και της γεωργίας, στην ε, μεταποίηση τροφίμων και στην ε, ε, στι πωλήσει λιανικών προϊόντων είναι πολύ περισσότερο αυτοί που επωφελούνται από τη φύση. Και από μια αρχική δουλειά που κάναμε είναι ότι είναι τριπλάσιοι οι δικαιούχοι σε σχέση με αυτό το οποίο φαίνεται στα στοιχεία του ΑΕΠ. Βλέποντας λοιπόν τον καινούριο πίνακα θα δούμε πραγματικά ποιος επωφελείται σε όλη την οικονομική αλυσίδα και αυτό θα μας δώσει κάποιες περισσότερες απαντήσεις στα ερωτήματα για τα ωφέλη. Τώρα κυρία Μακάβεν. Όχι τόσο για ερώτηση, αλλά για τα φαρμακευτικά, γιατί πριν ήμουν έξω για να τηλεφωνήσω. Συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο η Επιτροπή να ετοιμάσει έκθεση για την νομοθεσία όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν να κάνουν με το προϊόν για την ε, επαγρύπνηση, την φάρμακο επαγρύπνηση. Θα υπάρξει έκθεση από την Επιτροπή. Σας το λέω να το ξέρετε. Θα μπορούσα ίσως να γράψω στην Επιτροπή και να τη ρωτήσω ή να τη ζητήσω να έρθω σε επαφή μαζί σας για να βοηθήσετε. Ζητάμε και από τα κράτη-μέλη βέβαια να συνεργαστούν. Να φροντίσουμε να γίνει αυτό γιατί έχουμε νομική βάση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την ε, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που ήρθε σήμερα και είναι εδώ μαζί μας. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω από αυτό που είπε για τη νέα γεωργική πολιτική, την νέα ΚΑΠ, που, είναι, που έχει πάρα πολύ σημαντική θέση όσον αφορά το κοινό καλό. Μία γεωργία μπορεί να εξυπηρετήσει την προστασία του περιβάλλοντος και ε, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που είπε για τη χρήση του εδάφους και για την ε, διατήρηση του εδάφους και μάχη που δίδεται αυτή τη στιγμή, γιατί η οδηγία για την προστασία των εδαφών αυτή τη στιγμή κρατάται όμοιρος από κάποιες χώρες. Εγώ πιστεύω ότι αυτά εδώ δεν είναι βιώσιμα διότι ούτως ή άλλως το έδαφος είναι μια σπάνια, ένα σπάνιο αγαθό. Είναι μεν σταθερό, είναι εκεί, όμως έχει συνέπειες ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και δικαιολογούν απόλυτα μια πολιτική προστασίας και του υπεράσπισης του εδάφους. Κυρίως αναφορά τις νέες προκλήσεις που προέρχονται ακριβώς από τις κλιματικές αλλαγές. Από τις βροχές που είναι πολύ έντονες πλέον και επομένως η προσαρμογή η οποία πρέπει να γίνει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της επικράτειάς μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις το οποίο σημαίνει οι ικανότητες επεξεργασίας του εδάφους ε, και του νερού εκεί που βρέχει πολύ έτσι ώστε να ε, ε, εμπλουτιστούν εκ νέου οι υδροφόροι ορίζοντες και να περιορίσουμε τη διάβρωση του εδάφους όλα αυτά τα θέματα είναι απαραίτητα μεν, αλλά πανηρά δε. Γι' αυτό χρειάζεται να δούμε πώς θα γίνει επιτόπου η συντήρηση του εδάφους, αλλά και να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες που προσφέρουν και να νιώσουμε πηγές ενέργειες σε κάθε περιοχή. Για το έδαφος το πρόβλημα είναι τα κατάλοιπα, τα γεωργικά κατάλοιπα και τα δασικά κατάλοιπα επίσης. Θα πρέπει να γίνεται συντήρηση του δάσους, γιατί εκεί αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο κίνδυνο ε, πυρκαγιών. Έχουμε όμως ε, και τεράστιες ποσότητες βιομάζας που μπορούμε να πάρουμε από τα δάση. Γι' αυτό χρειάζεται μια συστηματική ενέργεια που θα γίνεται η συγκομιδή και η εκμετάλλευση της βιομάζας να αποτελεί, αποτελέσει ένα ουσιαστικό, ένα σημαντικό πόρο, γιατί με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουμε καλύτερα στην, προσαρμογή, στην αντιμετώπιση της στις συνέπειε των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει επομένως ε, να έχουμε μια συστηματική, μια καλή επεξεργασία και χρησιμοποίηση της ε, βιομάζας, αλλά και ε, διαχείριση των υδάτων, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατή πηγή υδατός με αποτελεσματικό τρόπο. γιατί κάθε, ε, κάθε, κάθε ποσότητα, οποιαδήποτε ποσότητα νερού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ε, συντηρούμε και διατηρούμε ε, το έδαφος. Όλα αυτά εμφανίζονται στην έκθεση, μια έκθεση την οποία πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Βιτόριο, ο καθηγητής κ. Κουλός. Thank you Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω εδώ και να σας μιλήσω, να απευθυνθώ σε σας. Όχι τόσο για να απαντήσω σε ερωτήσεις, όσο για να σας ενημερώσω, μια που είμαι παρόν στο Προεδρείο και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαι εδώ με τον κύριο Χολσμπεκ, τον συναδελφό μου. Έχω το προνόμιο να σας εκπροσωπώ από τότε που δημιουργήθηκε ο οργανισμός. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι η έκθεση, αυτή εδώ ειδικά η έκθεση, δεν είναι τόσο αισιόδοξη. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν φέρνει καλά νέα. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι άσπρα ή μαύρα, είναι συνήθως γκρι, σε διάφορες αποχρώσεις του γκρι. Ένα μοσαϊκό αποχρώσεων του γκρι. Αυτό που είναι καινούριο όμως και πρέπει να μας ικανοποιήσει εδώ στο Κοινοβούλιο είναι η φύση της έκθεσης. Ξεκινήσαμε με εκθέσεις που παρουσίαζαν την εικόνα με κάποιες επεξηγήσεις. Και έχουμε προχωρήσει τώρα σε εκθέσεις με ανάλυση, σύνθεση και σήμερα κάνουμε αξιολόγηση. Και προσπαθούμε όχι μόνο να καταλάβουμε διάφορα φαινόμενα βάσει των συμπτωμάτων τους, αλλά να εντοπίσουμε και τις αιτίες. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Δεν γνωρίζω βέβαια πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τα μέσα που έχει ο οργανισμός στη διάθεσή του. Και το θίγω αυτό, διότι η επιτυχία του οργανισμού και η καλή αυτή έκθεση δεν θα πρέπει να αποτελέσουν και παγίδα. Έχω την αίσθηση από τη συζήτηση, έτσι όπως διξάγεται εδώ σήμερα, ότι ίσως ζητήσουμε από τον οργανισμό υπερβολικά πολλά πράγματα συγχρόνως. Ζητάμε από τον οργανισμό ε, πολιτικές ε, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ζητάμε να απαντήσει στην Επιτροπή για πολιτικές που μερικές φορές δεν ε, είναι συνεκτικές μεταξύ τους και συγχρόνως ζητάμε από τον οργανισμό να βοηθήσουν τις χώρες να εφαρμόσουν τους κανόνες. Όλα αυτά είναι πάρα πολλά. Πιστεύω ότι ο οργανισμός προσπαθεί πραγματικά να το κάνει, βρίσκοντας μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα. Μην το ξεχνάμε αυτό όταν θα δώσουμε οδηγίες για το μελλοντικό έργο του οργανισμού. Έπειτα, όσο πιο πολύ εμβαθύνουμε στην ανάλυση, παρά την εξαίρετη βάση που έχουμε στην διάθεσή μας, παρόλα αυτά Όλα αυτά δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχνάμε ότι πρόκειται για οργανισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε στοιχεία από άλλους οργανισμούς και Ινστιτούτα. Και είναι κάτι το οποίο επιτυχώς το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τώρα όμως, εδώ και τώρα, είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να δώσει στον οργανισμό τα μέσα που χρειάζεται και συγχρόνως την εντολή που χρειάζεται με σαφήνεια. Διότι ζητούμε οργανισμούς που δίνουν στατιστικά δεδομένα και τα αναλύουν, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε την αξιολόγηση και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Αν όντω αυτός είναι ο ρόλος και το καθήκον που θέλουμε για την, ε, για τον οργανισμό περιβάλλοντος και θέλουμε αυτά, αυτές τις στατιστικές δηλαδή να ζητήσει από τις επιμέρους οργανώσεις. Αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι τώρα. Είναι πιστεύω πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε όπως προτάθηκε εδώ και νομίζω ότι ορθώς. Αν θέλουμε λοιπόν ο οργανισμός να καλύψει και να συνδυάσει περιβαλλοντικά στοιχεία με οικονομικά στατιστικά στοιχεία, με δημογραφικά, υγεία κλπ. Χρειαζόμαστε και περισσότερα χρήματα, αλλά και ευρύτερη εντολή για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Κάτι άλλο τώρα για το θεωρητικό σκέλος. Βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο αφηρημένου, το οποίο δεν γίνεται απαραίτητα κατανοητό από τις διάφορες αρχές. Και αυτό γιατί βασιζόμαστε σε έναν ενδιάμεσο κρίκο που θα δείξει στις περιφερειακές και τοπικές αρχές πώς μπορούν να συνδυάσουν τις διάφορες πολιτικές. Αν όμως το θέλουμε αυτό, τότε πρέπει να μας βοηθήσετε εσείς ζητώντας οικοδόμηση ικανοτήτων όχι μόνο σε τρίτες χώρες, αλλά και μέσα στην Ευρώπη, σε εθνικές και τοπικές αρχές. Χρειάζεται κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα. Εμείς μπαίνουμε σε μία περίοδο και σε ένα χώρο όπου οι πληροφορίες και η κατανόηση για να μας έρθουν ικανοποιητικά χρειάζεται κατάρτιση. Αλλιώς η επόμενη έκθεση δεν θα είναι τόσο αισιόδοξη. Αυτή την πρόγνωση κάνω εγώ. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο. Ξεκινήσαμε συζητώντας για τα πάντα και μην καταλαβαίνοντας τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Συνεπώς, βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό ο οργανισμός να έχει και την εντολή και τα μέσα που χρειάζεται και τις κατευθύνσεις που χρειάζεται για να κάνει περισσότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκούλο. Κυρία Μαγκλέιτ, θέλετε να καταλήξετε σε συμπεράσματα μετά από αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Και θα ήθελα να πω και προς τον κύριο Πρώτη ότι τα εδάφη θεωρούνται πολύτιμος πόρος. Το οικοσύστημα, γενικότερα αν το δούμε ως τμήμα του πώς οργανώνουμε τις συζητήσεις μας για την αποτελεσματικότητα, γιατί το έδαφος και η βιοπικιλότητα αλληλεμπλέκονται. Και έχετε δίκιο ότι στο πώς κατανοούμε τη σημασία των δασών ε, έχει εμποδιστεί από ε, τα προβλήματα που υπήρχαν με την οδηγία για τα εδάφη. Προσπαθούμε να είμαστε σε συνομιλία με τις διάφορες χώρες και μαζί με το πρόγραμμα GMS e θέλουμε να έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα μετά από 7 χρόνια που ήρθα στον οργανισμό, νομίζω ότι τελικά ε, βρήκαμε μια άκρη με τους γεωλόγους και υπογράψαμε μια συμφωνία ε, με όλες τις υπηρεσίες ε, στην Ευρώπη ώστε να απελευθερώσουν τους χάρτες τους και να τους διαθέσουν το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για το θέμα των δασών. Τα κατάλληλα πρέπει να εξεταστούν με μεγάλη προσοχή και δεν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε ένα πόρο και μόνο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Σημείωσα αυτά που είπε ο κύριος Κούλος και ένα τελευταίο σημείο για την επίπτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχουμε πιστικά δεδομένο ότι υπάρχει νομοθεσία ε, ε, στην οποία όλα τα κράτη ε, υπακούν, αλλά υπάρχει, υπάρχουν και άλλοι τομείς νομοθεσίας ε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εντάσσεται κατά διαφορετικό τρόπο γιατί υπάρχουν και θέματα ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να δούμε λοιπόν πού τίθενται οι φραγμοί και τι κάνει η νομοθεσία για να εντείνουμε την βιωσιμότητα και για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους πόρους και τι κάνουμε βάζοντας κάποια επίπεδα παραπάνω που τελικά στην αγορά δεν μας βοηθούν ή μπορεί και να λειτουργούν εναντίον μας γιατί μπορεί να έχουμε ένα πρότυπο ISO που εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και εγώ έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ευχαριστώ και τον Τζοκ και όλους τους συναδέλφους που είστε εδώ παρόντες ε, και ελπίζω να χαρείτε με την ανάγνωση της έκθεσης ε, όχι μόνο σε αυτά που σας παρουσιάσαμε εμείς σήμερα αλλά και το υπόλοιπο τμήμα του κειμένου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μακλέιντ. Νομίζω ότι όλοι εκτιμήσαμε την παρουσίασή σας. que nous, nous Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συζητήσουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση και τα δικαιώματα εκπομπών. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με προσώπους της Επιτροπής για το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Φιλίπ Φρανσουά. Μέχρι του έρθει ο κύριος Κράμερ. Κύριε Φρανσουά. Α, όχι, ήρθε, έρχεται και ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Φωνσουά από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα καταρχάς να ε, ζητήσω συγγνώμη, διότι η υπεύθυνη τη υπηρεσία μα ήθελε να έρθει σήμερα το απόγευμα εδώ, αλλά για λόγου υγεία δεν μπόρεσε να έρθει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόσκληση, για να περιορίσουμε την, για να παρουσιάσουμε το έργο τη Γενική Διεύθυνση ε, περιβάλλοντος για, τα, για τις συνέπειες ε, του εμπορίου των δικαιωμάτων εκπομπών για κάποιους συγκεκριμένους ρήπους ε, και τι γίνεται και με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Θέλω να σας δώσω κάποιες συγκεκριμένες, ε, κάποιες συγκεκριμένες στοιχεία και να σας δώσω και κάποια αποτελέσματα, αποτελέσματα των μελετών που έκανε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Καταρχάς να σας εξηγήσω γιατί η Επιτροπή μελέτησε την δυνατότητα να εφαρμόσει το εμπόριο δικαιωμάτων ε, για, τα, για, τις, για τις εκπομπές ε, ρήπων από τις, ε, τα άζωτα άζωτο ε, από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια υψηλή προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο ε, προσπαθούμε να βρούμε έναν αποτελεσματικό και όσον αφορά το κόστος τρόπο διαχείρισης των εκπομπών. Κάναμε μια μελέτη αντικτύπου μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της οδηγίας ε, του 2006 και 2007 και η μελέτη αυτή έδειξε ότι η εφαρμογή του εμπορίου δικαιωμάτων εκπομπών ε, σε αυτή, αυτούς τους δύο ρήπους μπορεί να περιορίσει το κόστος ε, της βιομηχανίας, ταυτόχρονα να έχει και μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά όμως, στο τέλος του 2007 καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα χρειαζόντουσαν περαιτέρω μελέτη και παρακολούθηση για να δούμε όλες αυτές τις πτυχές του συστήματος για το πού, πώς, θα έπρεπε να προσανατολιστούμε και πόσο θα έπρεπε να ε, ορίσουμε το, τα χρήματα, το, τα ποσά. Εξού και το 2007 δεν προχωρήσαμε. Όμως σε μια ανακοίνωση που συνόδευε την πρόταση αυτή δεσμευθήκαμε να εξετάσουμε περαιτέρω τα θέματα αυτά, να δούμε τι συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτό το ενδεχόμενο εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών και στην οικονομία και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι μελέτες αυτές βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και μας επέτρεψαν στο τελευταίο 1,5-2 χρόνο, χρόνια να κάνουμε μια μελέτη και μια αξιολόγηση και να συζητήσουμε με τους διάφορους εμπλεκομένους. Και τώρα βρισκόμαστε, όπως σας είπα, στο, στα, τελικά, στα τελικά στάδια ε, α, ε, συλλογής και αξιολόγησης των συγκροματικών πληροφοριών. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το οποίο μελετήσαμε δεν ε, είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα, ε, θα αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα command and control, θέλετε, στην ε, οδηγία για τους βιομηχανικούς ρήπους. Θα, θα αντικαταστήσουμε τις απαιτήσει της οδηγίας με αυτό το νέο εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών για τα διοξίδια του αζότου κτλ. Για να το για να ξεκαθαρίσω το θέματα, τα θέματα αυτά, ε, αυτό το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών για τα, ε, για το οξύδια του αζότου θα αντικαταστήσει αυτό το σύστημα το οποίο ήδη υπάρχει, θα, θα εφαρμόζεται σε συστήματα παρακολούθησης και αδειοδότησης των ε, βιομηχανικών καταστάσεων. Όμως όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της οδηγίας για, τις, για, την, για την οδηγία που αφορούν τις βιομηχανικές καταστάσεις θα παραμείνουν ενισχύ. Τώρα, για αυτές τις δύο μελέτες, να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες, σας είπα ότι έχουμε κάνει δύο μελέτες που ξεκίνησαν το 2009. Η πρώτη μελέτη ολοκληρώθηκε στα μέσα αυτής της χρονιάς και η δεύτερη μελέτη ε, ήταν ε, η συνέχεια αν θέλετε και τώρα βρίσκεται στα τελευταία στάδια. Η πρώτη μελέτη σε γενικές γραμμές εξέτασε τον, τις συνέπειες των, ε, κάποιου εμπορίου των δικαιωμάτων εκπομπών ε, στο περιβάλλον και στην οικονομία. Ε, εξετάσαμε 20 πιθανά σενάρια με διαφορετικές παραμέτρους στο εμπόριο των δικαιωμάτων. Η δεύτερη μελέτη είχε σαν στόχο να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες, να κάνει μια περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών συνεπειών π.χ. ανταγωνισμό, εσωτερική αγορά, διεθνή ανταγωνιστικότητα, ε, δημιουργία θέσεων απασχόληση. Τα αποτελέσματα τη πρώτη μελέτη που τα έχουμε στη διάθεσή μα από τα μέσα αυτή τη χρονιά ε, μα λένε ότι το εμπόριο των δικαιωμάτων αυτού του δύο ρήπου ε, θα μπορούσε να περιορίσει τι εκπομπέ διοξιδίων του αζότου και του θείου ε, θα περιοριστούν και με περιορισμένο κόστος για την ε, κοινωνία. Δηλαδή θα έχουμε και χαμηλότερες εκπομπές από ό,τι θα είχαμε με, αν εφαρμοζόταν ως ε, έχει η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και, πολύ με, και με χαμηλότερο κόστος. Η άλλη μελέτη λέει ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα, αρκεί βέβαια να εφαρμοστούν κάποιες ε, συγκεκριμένες ρήτρες, ε, λόγω όμως της, των περιορισμένων εργαλείων που είχαμε στη διάθεσή μας, παρόλο που χρησιμοποιήσαμε τα καλύτερα ποιοτικά εργαλεία, ε, χρειαζόμαστε, πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια επιφύλαξη αν θέλετε. Τώρα, ένα άλλο συμπέρασμα σημαντικό για τις πρώτες μελέτες είναι το, το οικονομικό κόστος και οι εξοικονομήσεις από αυτό το ενδεχόμενο εμπόριο των δικαιωμάτων θα, εξαρτηθεί, θα εξαρτηθούν από, τις, από το πώς θα εφαρμοστεί το σύστημα και ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες, ε, δηλαδή πώς θα κατανεμηθούν ε, η, τα χρήματα, ε, ε, εάν θα γίνει μέσα πλαίσια δημοπρασίας, ε, εάν θα ορίσουμε εμείς συγκεκριμένα ποσά κτλ. Όλα αυτά επιβεβαίωσαν πόσο σημαντική, με σημαντικό είναι το σύστημα κατανομής και θα πρέπει να δούμε τα έσοδα από τις δημοπρασίες πώς θα αποφασιστούν, πώς θα, χρησιμοποιηθούν κτλ. Πάντως η δεύτερη μελέτη απέδειξε ότι για όλη την Ένωση ε, το, η εφαρμογή αυτού του συστήματος ε, ε, σε κάποιους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν θα έχει μεγάλη επιρροή. Επίσης θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία και στις συζητήσεις για την εφαρμογή αυτού του εμπορίου των δικαιωμάτων εκπομπών ε, οξυδίων του αζότου και του θείου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα σχόλια από τους εμπλεκομένους. Μας βοήθησαν τα σχόλιά τους για να διαμορφώσουμε τη, τη συνολική μας εικόνα και καλωσορίζουμε επίσης και το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά. Κυρίως ε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα την αλληλεπίδραση του εμπορίου των δικαιωμάτων εκπομπών και τις ε, νομοθεσία, συγκεκριμένα την οδηγία υγεία για τις βιομηχανικέ εκπομπές. Επίση, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα ότι τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο τη ανάλυση. Οι δύο μελέτε είναι στο τελευταίο, τελευταία φάση ολοκλήρωσή του και μία απόφαση για το κατά πόσο θα προχωρήσουμε για το, για το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών οξυδίων του αζότου και του θείου θα ληφθεί στο άμεσο μέλλον. Πρέπει να έχουμε όμω μια σαφέστερη εικόνα για τι δυνατότητε και για του περιορισμού που ένα τέτοιο εμπόριο ε, θα είχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλησπέρα. Ε, ζήτησα το λόγο γιατί είμαι εισηγητής για την ε, αναθεώρηση της οδηγίας IPPC για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρήπανσης και έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το έργο μας και παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή επεξεργάζεται ένα νέο εργαλείο για την ατμοσφαιρική ρήπανση στην Ευρώπη και υπάρχουν διάφορα κέρια ερωτήματα. Ακούσαμε και τις δηλώσεις της Επιτροπής, τις οποίες ε, κατανοήσαμε ε, ως ότι δεν πρόκειται να υποβάλει μια νέα πρόταση, αλλά είναι σε μια φάση που κάνει μελέτες ε, και αξιολόγηση επιπτώσεων για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των μέσων που θα επιλεγούν. Αυτό το οποίο συχνά ε, λέμε είναι ότι είμαστε πολύ διστακτικοί και πολύ κριτικοί έναντι των ε, όσων μας λέει η Επιτροπή. Διότι υπάρχει μια οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές που δεν είναι επιτυχημένη μεν, αλλά υπάρχει ένα νομοθετικό μέσο. Αυτή η οδηγία τώρα τροποποιείται και υπάρχει μια σημαντική πρόοδος, επιτυχία θα έλεγα, ε, στο ότι η δυνατότητα ε, απόκλησης από την ε, βέλτιστη τεχνική είναι κάτι το οποίο αναφέρεται. Αυτό το νέο διατυπωθέν άρθρο θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη και να δούμε πώς θα αποβεί στην πράξη. Πρέπει να βρούμε διατυπώσεις για να δούμε ε, τι θα γίνει συγκεκριμένα στην πράξη, στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ε, από όσα έχω ακούσει από πολλά κράτη-μέλη και μάλιστα από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν μεταφέρει σε εθνικό δίκαιο με επιτυχία την οδηγία IPPC, ε, βλέπω ότι θα περιμένουν να δουν πώς θα πάει αυτό το νέο νομικό μέσο. Δηλαδή θα δουν αν το μέσο το οποίο ήδη βρίσκεται σε λειτουργία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και νομίζω ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να σκεφτούμε ένα σύστημα με οριακές τιμές και να αντικαταστήσουμε με το εμπόριο εκπομπών. Γιατί στην πρακτική ε, μετατροπή θα υπάρξουν προβλήματα και νομίζω ότι δεν το φαντάζεστε καν τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ε, θέτω το ερώτημα αυτό και σε μένα και άμεσα στην Επιτροπή. Πώς λειτουργεί ένα σύστημα όπου ε, ορίζονται οριακές τιμέ για, τη βιομηχανή, για βιομηχανικές εγκαταστάσεις επί τη βάση του BVT και πώς λειτουργεί ένα σύστημα στο οποίο υπάρχουν οριακές τιμές ε, για μεγάλες εγκαταστάσεις ε, καύσης παράλληλα με το εμπόριο εκπομπών. Δεν αποφασίζουμε το πώς θα λειτουργεί και τι κάνουμε στα κράτη-μέλη όπου μέχρι τώρα έχει προχωρήσει νομοθεσία για ε, τις εκπομπές και υπάρχουν συστήματα σε λειτουργία και επιτυχημένα συστήματα και σιγά σιγά είπαμε ότι αλλάζουν και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σύστημα λοιπόν το οποίο λειτουργεί, γιατί θέλουμε να το αντικαταστήσουμε με το εμπόριο εκπομπών. Ή νομίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα σταματήσουν να ισχύουν οι εθνικοί νόμοι για να ισχύει ξαφνικά το εμπόριο εκπομπών. Πρέπει βέβαια από την άλλη πλευρά να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές ε, του κόσμου που υπάρχουν θετικές εμπειρίες με το εμπόριο εκπομπών για τους ατμοσφαιρικούς ρήπους. Και είναι επιτυχημένα τα συστήματα κυρίως διότι είναι οργανωμένα τοπικά και περιφερειακά. Από ό,τι καταλαβαίνω από την Επιτροπή μιλάει για ένα σύστημα εμπορίου εκπομπών για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ παραπέμπω ε, στο εμπόριο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος που δεν καταφέραμε ε, να έχουμε μια δίκαιη κατανομή μεταξύ κρατών μελών και σημαντικών ε, εταίρων παράλληλα. Γιατί λοιπόν θα λειτουργήσει τώρα αυτό το σύστημα για τους ατμοσφαιρικούς ρήπους καλύτερα. Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που είναι ήδη πολύ προχωρημένα στα θέματα αυτά. Είναι, υπάρχουν κράτη-μέλη όπου δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό το τομέα. Και θα βάλουμε κάποιο ανώτατο όριο για τα οξύδια του αζότου και παράλληλα θα προσπαθήσουμε να υποχρεώσουμε τα, τα κράτη-μέλη σε ακόμη περισσότερες αλλαγές ε, και όχι ανάλογα με το τι έχουν επιτύχει μέχρι τώρα. Η Επιτροπή πάντοτε τονίζει πόσο σημαντική είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την οδηγία IPPC. Και ε, ξέρουμε ότι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις πάντοτε υπάρχουν ρήποι, πάντοτε υπάρχουν εκπομπές ε, και η ατμοσφαιρική ρήπη είναι ένας από τους ρήπους, ένα από τα επιβλαβή στοιχεία. Και όταν μιλάμε για ολοκληρωμένη προσέγγιση, σημαίνει ότι όταν αφήνουμε κάτι να είναι υψηλότερο, κάτι άλλο θα είναι χαμηλότερο και αντιστρόφως. Το εμπόριο εκπομπών ε, για τους ατμοσφαιρικούς ρήπους ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβαδίζει με την ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση. Είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα που ανέφερα. Θα πρέπει η Επιτροπή πολύ προσεκτικά να σταθμίσει την σημασία μιας αλλαγής του συστήματος στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και όχι να γίνει κάτι από τη μία στιγμή στην άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο. Αρσένης, Βίζας, Ζαμπέρ, Λίντα Μακάβεν. Κλείνει εδώ ο κατάλογος. Και εσείς. Γι' αυτό το σημείο. Ή για το επόμενο. Ή για το σημείο 7 του 23. Το 7 ήταν για αύριο το πρωί που έχει να κάνει επίση με τις άδειες. Και είναι και ο κύριος Κυλακάκης, δεν είναι, που είσαστε συγκητές μαζί για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι. Ωραία, δύο λεπτό καθένα. Σύμφωνοι. Γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα ακόμα να εξετάσουμε. Οπότε, Κρήτον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή. Έχει κάποιες τιμές ε, στο μυαλό της ε, για τα οξύδια του αζότου. Τι τιμές έχει υπόψη της για τα αέρια του και για το διοξίδιο του άνθρακα και για το οξίδια του αζότου και για το μονοξίδιο του αζότου. Και για να δούμε και πιο πέρα λίγο τα πράγματα. Ξέρουμε ότι στο σύστημα αυτό εμπορία δικαιωμάτων υπάρχουν ελλείψεις και ασφάλματα. Το 2009 για παράδειγμα. Πώς θα αποφύγουμε τέτοιες αποτυχίες αν συμπεριλάβουμε και τα οξύδια του αζότου και το διοξίδιο του θείου. Άνια Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παράλληλα με την ερώτηση που έκανε ο συνάδελφο Κράμερ, θα ήθελα να πω ότι οι βιομηχανικέ εκπομπέ του ανοξιδίου, του αζώτου και του διοξιδίου του θείου έχουν μειωθεί τι τελευταίε δεκαετίε και αναμένει κανεί ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. και η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές ε, που πρόσφατα εγκρίναμε προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. «47% και 66% για το οξύδιο του αζότου και το διοξίδιο του θείου είναι οι μειώσεις τις οποίες ε, ε, ελπίζουμε και υπάρχουν ε, πολλοί φορείς και πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που έχουν εκφράσει ανησυχία και για την ε, αποτελεσματικότητα έναντι του κόστους και για το εφικτό του εμπορίου εκπομπών οξυδίων του αζότου. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή τι περιμένει από αυτό το νέο σύστημα ε, εμπορίου εκπομπών, τι προστιθέμενη αξία περιμένει η Επιτροπή ε, από την αλλαγή από ένα σταθερό σύστημα τιμών σε ένα σύστημα εμπορίου και τι επιπλέον επιβαρύνσεις θα υπάρχουν ενδεχομένως δεν θα υπάρχει αποτελεσματική μείωση των εκπομπών. Γιατί να αλλάξουμε λοιπόν ένα σύστημα που είναι επιτυχημένο, που αποδεδειγμένα έχει οδηγήσει σε μείωση ε, των εκπομπών. Δεν μου είναι σαφές και γι' αυτό θα ήθελα ε, να ακούσω τι έχει να πει η Επιτροπή και συμφωνώ με όσα είπε ο συνάδελφος Κράμερ. Ε, ε, ο Ορέστη Ρώση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο διευκρινήσεις. Καταρχάς ε, ανησυχώ για τον τρόπο πώς ε, γίνεται η, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των, των δικαιωμάτων εκπομπών. Διότι δεν θέλουμε να γίνουν στον τομέα αυτό κερδοσκοπικές κινήσεις. Και θέλουμε να ξέρουμε τι, προτίθεται, τι προτιθέμεθα να κάνουμε έτσι ώστε να μην ε, υπάρχει ένα είδος χρηματιστηρίου αν θέλετε όλων αυτών των ε, εκπομπών. Αυτό θα με ανησυχούσε ιδιαίτερα ε, αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση ούτως ή άλλως και δυσκολευόμαστε να την ε, ξεπεράσουμε. Επίσης, πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις επιλογές των κρατών μελών, διότι μιλάμε για 50% ε, χρήματα τα οποία προέρχονται από τις ε, δημοπρασίες και τα χρήματα αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν τα κράτη για, την, για το περιβάλλον, κλιματολογικές αλλαγές, περιβαλλοντική προστασία κτλ. Και το υπόλοιπο 50% θα το καθορίσουν τα κράτη-μέλη πώς θα το χρησιμοποιήσουν και Επομένως, θα πρέπει απλώς και μόνο να ενημερώσουν την Κομισιό για τις ε, αποφάσεις τους. Ή απλώς το κείμενο εδώ δεν μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες ε, και δεν λέει ε, η Κομισιόν τι θα το κάνει. Αυτό το 50% που είναι σημαντικό ποσό το κράτος μέλος θα το κάνει ό,τι θέλει χωρίς να δίνει κανένα λόγο στην Κομισιό ή πώς παρεμβαίνει η Κομισιόν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Παρακαλώ, εσείς. Θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την εμπειρία που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα από το σύστημα αυτό. Είδαμε στο CDM προβλήματα με τον μηχανισμό αυτών ε, εμπορίας δικαιωμάτων, αλλά και αλλού και σε άλλες περιπτώσεις. Σήμερα έχω μια απάντηση από την Επιτροπή. Για πρώτη φορά θα δει το ποιος είναι υπεύθυνο για τα θέματα αριθμίας ε, ή ατασταλιών που διαπιστώνονται στην αγορά. Ποιος ευθύνεται. Έχω και ερωτήσεις για ένα σύστημα που είναι φτιαγμένο για την εμπορία. Το διοξίδιο του άνθρακα, όπως καταλαβαίνετε, ε, δεν έχει σύνορα. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση για εμπορία. Σε περιπτώσεις τώρα οξυδίων του θείου και του αζότου υπάρχει και τοπικός παράγοντας. Έχετε δηλαδή πολύ περισσότερο τοπικά τις εκπομπές από ό,τι έχετε με το διοξίδιο του άνθρακα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μπαίνοντα σε αυτή την περιπέτεια. Πρέπει να δούμε και άλλους τρόπους χειρισμού πριν αποφασίσουμε για το σύστημα εμπορίου δικαιωμάτων εκπομπών. Αν μη τι άλλο, Πρέπει να βρούμε λύσεις στα προβλήματα του συστήματος εμπορίας πριν βάλουμε και άλλα πράγματα εκεί μέσα. Ο κύριος Κρότε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λαμβάνοντας υπόψη το εμπόριο για τις αεροπορικές μεταφορές είχαμε ε, συζητήσει και ε, με πολλές συζητήσεις με την Επιτροπή ε, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα και είχε πει η Επιτροπή ότι κάτι θα μας παρουσίαζε για τα οξύδια του αζότου στις αερομεταφορές και μου κάνουν εντύπωση αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Κράμερ για τις βιομηχανικές εκπομπές. Θα ήθελα να μας δίνατε μια απάντηση ε, για το τι έχει γίνει σε σχέση με την πρόταση εκείνη. Τώρα όσον αφορά το CDM, το Μηχανισμό Πρωτοκόλλου Καθαρής Ανάπτυξης που ανέφερε και ο συνάδελφος. Έχουμε τα πιστοποιητικά και το πρόγραμμα για το 23 Ε, ξέρουμε ότι το, το CDM, ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης, είναι καλό μέσο, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το διεθνές και γι' αυτό θα ήθελα μια δήλωση της Επιτροπής τι, μπορεί, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην υπάρχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για ορισμένε εταιρείε και για να κλείσουμε το κενό το οποίο υπάρχει στον τομέα του CDM. Ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω τώρα από την Επιτροπή να απαντήσει όσο πιο σύντομα μπορείτε. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Με αυτές που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τις δράσεις για το περιβάλλον θα τις αφήσω για τους συναδέρφους από το περιβάλλον. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό λοιπόν εκ με ένα σύστημα που βασίζεται στις τιμές εκπομπών. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, ότι αυτό που κοιτάξαμε, αυτό που μελετήσαμε ήταν ένα σύστημα που θα αντικαταστήσει την απέτηση για τις οριακές τιμές, για τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το ε, σύστημα εμπορίου εκπομπών. Δεν είναι επιπλέον. Όμως, όπως επίσης είπα στην αρχή, μπορεί να χρειαστεί να κρατήσουμε ή να αναπτύξουμε κάποιες ε, ρήτρε ασφάλειας κατά κάποιο τρόπο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και δυνατότητες που ίσως προκύψουν τοπικά με την εισαγωγή του εμπορίου αυτού των δικαιωμάτων εκπομπών. Οι τοπικές ε, εκπομπές είναι ένα ενισχυτικό στοιχείο και γι' αυτό θα έπρεπε όντως να το κοιτάξουμε περισσότερο γιατί το τρέχον μοντέλο δεν μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε απόλυτα αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα το εύρος. Σκεφτήκαμε ένα σύστημα πανευρωπαϊκό, αλλά βέβαια κάποια σενάρια και κάποιες μελέτες ήταν πιο τοπικές, δηλαδή περιφερειακές πιο σωστά, περιλαμβάνοντας λίγες χώρες μόνο. Ευθύ εξ αρχή είπαμε ότι το σύστημα κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να βασίζεται σε κανόνες που να ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύουμε ότι όσο ευρύτερο είναι το σύστημα εμπορίας, τόσο πιο αποτελεσματικό οικονομικά θα είναι. Γιατί θα υπάρξουν περισσότερα δικαιώματα για εμπορία. Όσον αφορά τώρα τα διαφορετικά σημεία κίνησης, Νομίζω ότι εδώ πολύ σημαντικό είναι, για να μην πληγεί αυτός που πιο νωρίς ξεκινάει, Σωστό είναι λοιπόν να κοιτάξουμε συστήματα τα οποία μπορούν να πετύχουν τα ίδια επίπεδα φιλοδοξιών σαν αυτά που έχουμε στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές όπου εκεί όσον αφορά τις επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος είχαμε πάντα τη, ως σημεία αναφορά στις μελέτες που έχουν γίνει και όταν μιλάμε για δυνητικό εμπόριο πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σενάριο με σημεία αναφοράς. Όποιοι και αν προτιμηθεί, αν μη τι άλλο, πρέπει να έχει το ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικών φιλοδοξιών. Συνεπώς, οι εκπομπές πρέπει να βασιστούν στην εφαρμογή του BET, της ε, βέλτιστης δηλαδή διαθέσιμης τεχνολογίας και αυτό θα καθορίσει τις φιλοδοξίες μας για το περιβάλλον. Δεν έχουμε συγκεκριμένη τιμή ή ελάχιστη τιμή για τα δικαιώματα. Για την ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις βιομηχανικές εκπομπές. Εδώ πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι για τις άλλες περιπτώσεις πριν του θείου και του αζότου διατηρούνται οι ίδιες συνθήκες. Οι οριακές τιμές δηλαδή, οι άλλοι περιορισμοί που ήδη υπάρχουν. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η εμπορία δικαιωμάτων θα αλλάξει κάπως το τη σημερινή κατάσταση. Κοιτάμε λοιπόν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των μελετών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και τις αντιδράσεις που έχουν φτάσει σε εμά από τους ενδιαφερόμενους και θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας πριν καταλήξουμε σε απόφαση για το ναι ή όχι θα προχωρήσουμε με ένα τέτοιο σύστημα. Όσον αφορά την ερώτηση ποια είναι προστιθέμενη αξία του συστήματος ή ποια πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι αυτή. Ευθύ εξ αρχή είπαμε ότι προσπαθούμε να βρούμε ένα σύστημα που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ε, αποτελεσματικότητα κόστους, αλλά με το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας μας για το περιβάλλον. Αν υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό ήταν και το νήμα που ακολουθήσαμε και εκπονήσαμε τα διάφορα σενάρια. Αυτό. Τελειώσατε, λέει ο Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Προτείνω, μια και πρόκειται για το ίδιο θέματα, ή τουλάχιστον προσεγγίζει με αυτό εδώ, αύριο το πρωί, στο 23, στο σημείο 23, στο σημείο 7, που έχει να κάνει με, την, με το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων που συνεισφέρουν στην ατμόσφαιρα, ε, στην ατμοσφαιρική ε, συνάδοση θερμοκρασία, συγγνώμη, και δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε σχέση με τις ερωτήσεις ε, που ετέθησαν για το, για το εμπόριο δικαιωμάτων κάποιων ρήπων, η, το Συμβούλιο έδωσε στην Κομισιό αρμοδιότητες ε, να εφαρμόσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιων διατάξεων ε, από το 2013. Η Κομισιό προτίθεται να υποβάλει μία πρόταση, την οποία κάναμε, για τα HFC και για κάποια συγκεκριμένα οξέα που θα ισχύσουν από, την, από το 2013. Αφορούν 23, 23 ε, ουσίες. Η πλήρης μελέτη του αντικτύπων και ένα κείμενο ερωτήσεων-απαντήσεων δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα και θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις ε, των βουλευτών. Όπως είπε και η Επίτροπος Χιντεγκάρκα, δεν ε, θέλουμε να έχουμε λιγότερες πιστώσεις. Ε, ίσα ίσα υποστηρίζουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις αλλαγές του κλίματος και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν και σημαντικές συνέπειες στην τιμή του κοινοτικού άνθρακα. Τώρα, όσον αφορά την αγορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στο πακέτο ενέργειας και περιβάλλοντος ζήτησε να συμπεριληφθεί και μία έκθεση που να αφορά την αγορά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο, περισσότερο στο άρθρο 12 της οδηγίας. Προετοιμάζουμε μία ανακοίνωση για το θέμα αυτό που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο τους επόμενους δύο μήνες. Τώρα, όσον αφορά τις ε, τιμές στόχου, δεν υπάρχει, έχουμε τιμή στόχου μέσα στα πλαίσια του, EU, του ETS, του, του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών δηλαδή. Θέλουμε να πετύχουμε τους καλύτερους δυνατούς στόχους με το χαμηλότερο κόστος. Και λόγω της ύφεση ε, πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερα να έχουμε μια δέσμευση στο 30% των, της μείωσης. το μεγαλύτερο κομμάτι των ε, εσόδων από τις δημοπρασίες, το 50% δηλαδή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν ε, τις ε, αλλαγές του, του, κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή είναι μια δέσμευση την οποία να έχει αναλάβει το Συμβούλιο και θα πρέπει και εμείς και το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί ότι όντως τα κράτη-μέλη θα το θα εφαρμόσουν την υποχρέωση αυτή για την αεροπορία. Η υποχρέωση είναι 100% και για το υπόλοιπο 50% δεν υπάρχει ε, υποχρέωση των κρατών μελών. Τώρα όσον αφορά τις εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου από τα αεροπλάνα. Υπάρχουν δεσμεύσεις ε, και τις σας θυμίζω όταν υιοθετήσαμε αυτή την νομοθεσία η Κομισιόν και οι υπηρεσίες μας ε, εργάζονται έτσι ώστε οι, στις αεροπορικές μεταφορές να έχουμε πλήρη εφαρμογή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Κύριο, κύριο Σκυλακάκης και μετά κύριο Ζαρμπάντη. Θα, να είσαστε πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιό γιατί ακριβώς προχώρησε και προχώρησε γρήγορα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για τα θέματα αυτά. Ήθελα επίσης να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι όταν έχουμε απόδοση κεφαλαίου μιας, ε, ε, των, επενδύσεων σε 10, κατά 10%, σύμφωνα με τη μελέτη της Κομισιόν είναι εφταπλάσια τα αποτελέσματα. Επομένως αυτό το οποίο λέγαμε ήταν, είναι απόλυτα σωστό και αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις ότι τα συστήματα αυτά ε, καταστροφή του αερίου του HFC 23 έχουν ε, μας έχουν επιτρέψει να βγάλουμε πάρα πολλά χρήματα, διότι έχει γίνει απόδοση της επένδυσης πλήρης και θα πρέπει να δούμε το Κοινοβούλιο τι θα κάνει μέχρι το τέλος του 2012. Η δουλειά έχει κάνει την δουλειά, την Κομισιόν έχει κάνει τη δουλειά της, άρα εμείς σαν Κοινοβούλιο θα πρέπει να μιλήσουμε στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ζαμπράντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Όπως και ο συνάδελφος ο κ. Σκυλακάκης είπε, χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την κίνηση της Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ένα παράθυρο δύο ετών στο σύστημα και προσπαθώ να βρω τρόπο να το κλείσουμε αυτό το παραθυράκι, αυτό το κενό να το κλείσουμε. Ένας τρόπος και θα ήταν να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις μας, πράγμα το οποίο εγώ ήδη κάνω στη χώρα μου. Άλλος τρόπος θα ήταν να το συζητήσει η Επιτροπή Παραδείγματος Χάρη με την Business Europe να το συζητήσει μαζί τους, διότι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ένα παραθυράκι στην τρέχουσα νομοθεσία που δεν είχε την πρόθεση να έχει τέτοιες παράπλευρες ενέργειες και θα πρέπει να είναι πρόθυμη η βιομηχανία να αναλάβει μια τέτοια συμφωνία, να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις να μην μπουν σε αυτό το πρόγραμμα που επιτρέπει το παραθυράκι για τους ε, υδροφεράνθρακες 23. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να κάνει μια τέτοια κίνηση. Μια σύντομη απάντηση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Από τότε που τον Αύγουστο η Επίτροπο Χέντεγκαρντ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μια πρόταση επιτροπή, λάβαμε πολλά στοιχεία και πολλέ πληροφορίε από του εμπλεκομένου και από την Business Europe και το βάλαμε και στην ιστοσελίδα τη Επιτροπή στο πνεύμα τη διαφάνεια. Η Business Europe καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι υπέρμαχο τη πρόταση τη Επιτροπή. Αναμένεται λοιπόν ότι ο διάλογο θα συνεχιστεί. Η Επιτροπή έκανε μια πρόταση που θα ισχύσει από τη, συντομ, τη συντομότερη δυνατή στιγμή, πριν από τον Ιανουάριο του 2013, είναι κάτι που πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και δεν μπορεί να το επιβάλλει η Επιτροπή. Πάντως πριν από τον Ιανουάριο του 2013. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προτείνω να περάσουμε στο τελευταίο θέμα, το οποίο είναι η ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα, προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομική πόρη για μια βιώσιμη Ευρώπη μετά το 2013. Θα ήθελα να δώσω λόγο στον κύριο Ζεμπράντι, ο οποίος είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε κρατήσει το πιο καλό για το τέλος, ε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έχουν παραμείνει στην αίθουσα πάντως πόσο σημασία έχουν οι νέες δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Πολύ μεγάλη, το ξέρουμε. Μιλάμε για τη δημοσιονομική περίοδο μέχρι το 2020. Έχουμε διαπιστώσει ότι είναι κάπως στατικό τελευταία το σύστημα. Το 2010 όμως θέλουμε να έχουμε το πλαίσιο για μέχρι το 2020. Ήδη είχαμε το πενταετές σχέδιο, αλλά από εδώ και πέρα θέλουμε να έχουμε δεκαετές πλαίσιο. Τι σημαίνει το σύστημα. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ξοδεύουμε χρήματα τα οποία αποφάσισε η Ευρώπη το 2005 να ξοδέψει. Θα πρέπει, αυτό είχε γίνει επί Τόνι Μπλερ. Θα πρέπει λίγο να νεωθεί όμως το πράγμα. Το 2005 αποφασίσαμε σήμερα και μέχρι το 2013 πώς θα δαπανάμε τα χρήματά μας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές που είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, να δούμε τι θα συμφωνήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ήδη δυσκολευόμαστε για το 2011. Φανταστείτε για πιο μακριά. Στην έκθεσή μου που υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Λυπάμαι. Μου είπανε 1500 χτυπήματα έπρεπε να είναι η έκθεσή μου και όχι παραπάνω. Εγώ είχα βάλει και παραπάνω πράγματα, αλλά περιορίζομαι, βλέπετε, από τους κανόνες. Με το όνομά μου είναι και παραπάνω, μάλιστα, ξεπερνάω. Έβαλα λοιπόν τις προτεραιότητές μας. Ζητάω όμως εσείς να με βοηθήσετε για τη συνέχεια, για να διευρύνουμε κάπως ε, το κείμενο ή να το κάνουμε ακριβέστερο. Πώς μπορεί να επηρεάσει η έκθεση αυτή τώρα, η γνωμοδότηση μάλλον αυτή, την τελική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δημοσιονομικές Πρόπτικες, που ετοιμάζει ο κύριος ε, Δερίγα, ο κύριος Γκαρίγα. Εμείς έχουμε αυτήν την ε, έκθεση, υπάρχει γνωμοδότηση εκτός από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και από άλλες επιτροπές, η κυρία Χάουκ ε, και, η κυρία Μπάσχακ επίσης βοηθούν με την εκπόνηση της γνωμοδότησης αυτής της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες για την κάθε γραμμή στη γνωμοδότησή μου, αλλά κυρίως να μιλήσουμε για το όραμα που έχουμε για το μέλλον όσον αφορά την Ευρώπη. Και αυτό το όραμα να μπει στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν το καταφέρουμε αυτό, αυτό θα είναι μεγάλο επίτευγμα. Ακούσαμε σήμερα και την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ότι λείπει συνοχή πολλές φορές. Δύο είναι οι άξονες που ακολουθώ εγώ. Πολύ σημαντικό είναι η περίληψη του παράγοντα περιβάλλον στις άλλες πολιτικές. Όταν μιλάμε για την μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής, ελευτικής πολιτικής κλπ. κλπ το μήνυμα αυτό χάνεται. Εγώ θα ήθελα αυτό το μήνυμα να είναι και πάλι παρόν. Να συμπεριλαμβάνεται λοιπόν ο παράγοντας περιβάλλον και στους άλλους τομείς. Και να υπάρχουν και χρήματα γι' αυτό. Αντί να υπάρχουν χρήματα για να καταστρέφουμε το περιβάλλον. Και στην Αγγόγια για την βιοπικιλότητα αναφέρθηκε αυτό στους στόχους μας. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο κινούμε είναι αυτό που είπε ο Bill Clinton, economy stupid. Δηλαδή, να έχουμε μια πολιτική η οποία να έχει νόημα για το περιβάλλον. Πρέπει να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον. Αυτές να ενισχύουμε οικονομικά. Ας δούμε τι γίνεται και αλλού στον κόσμο με τα διπλώματα έβρεση τεχνίας για την πράσινη τεχνολογία είχαμε πει ότι η Ευρώπη θα πρωτοστατήσει στις, ε, στα φτηνά διπλώματα ευρεσιτεχνίες όταν πρόκειται για πράσινη τεχνολογία. Αλλά τελικά και εδώ η Κίνα έχει το πάνω χέρι. Αν δεν φροντίσουμε γι' αυτό περισσότερο, θα βρεθούμε πολύ πίσω. Πιστεύω λοιπόν ότι θα βρούμε δυσκολίες. Γιατί θα λείπουν τα ορυκτά. Και εδώ πάλι είναι η Κίνα που πρωτοστατεί όσον αφορά τον ορυκτό πλούτο. Θα είναι πιο ακριβώς ο ορυκτός πλούτος και αυτό θα μας πλήξει εμά. Έπειτα υπάρχουν τα λεγόμενα σπάνια μέταλλα τα οποία βρίσκονται ω επιτοπλίστων στην Κίνα. Και από τα 14 ορυκτά που είναι ζωτική σημασία για το μέλλον, η Ευρώπη δεν διαθέτει κανένα. Ο δεύτερος λόγος είναι η περιβαλλοντική νομοθεσία που όντως πρέπει να είναι τέτοια που να μας βοηθήσει να προχωράμε με βιώσιμη ανάπτυξη. Η Unilever είπε ότι το 2020 θέλει να είναι 100% βιώσιμη επιχείρηση. Αυτό έχει να κάνει και με την νομοθεσία αλλά και με την δύναμη αγοράς που διαθέτει ο καταναλωτής. Γιατί η το είπε αυτό. Αλλά είδατε τι γίνεται τώρα με το φινικέλαιο, για παράδειγμα, που κατέληξε σε μποϊκότ. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία γύρω από τα οποία κινείται η γνωμοδότησή μου. Και θα ήθελα να συμπεριληφθούν στην έκθεση του Κοινοβουλίου για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Οι δημοσιονομικές προοπτικές όμως είναι χρήμα, μιλούν για χρήμα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός στην Ευρώπη για το περιβάλλον είναι πάρα πολύ χαμηλός. 450 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ λίγο. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα αν δείτε τι θέλουμε να πετύχουμε. Γι' αυτό και γίνονται πολύ λίγα. Τα κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισαν ότι μόνο για το Natura 2000 χρειαζόμαστε 5,8 δισεκατομμύρια. Στην Κοπεχάγη πολλές υποσχέσεις ακούσαμε για τα δάση και ότι χρειάζονται 18 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστια τα ποσά αυτά. Και δεν θα τα βρούμε όλα αυτά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Χρειάζονται χρήματα όχι μόνο από το δημόσιο τομέα, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα για να τα καταφέρουμε. Τέτοια ποσά συνειδητά δεν τα αναφέρω στη γνωμοδότησή μου. Αυτό όμως που λέω είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε η Ευρώπη να είναι σε θέση να έχει επαρκείς πόρους στη διαθεσή της για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μας, τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας όσον αφορά το περιβάλλον. Κυρία Πρόεδρε, περιμένω με μεγάλη περιέργεια τις αντιδράσεις των συναδέρφων. Όπως είπα, αυτή η γνωμοδότηση αποτελεί ένα μόνο στοιχείο όσον αφορά το περιβάλλον που ελπίζω να συμπεριληφθεί στην έκθεση Γκαρίγκα του Κοινοβουλίου. Με έχει βοηθήσει πολύ η κυρία Χαουγ και θέλω να την ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως. Περιμένω τις αντιδράσεις σας τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Dan. Øh, øh, Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή μας για αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις και για όλη τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Φτάνει πολύ καλά η στιγμή συζήτησης αυτής της έκθεσης, ακριβώς μετά την παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Μακλέιντ για ε, την κατάσταση του περιβάλλοντος για το 2010. Πολλά από τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε να μπορέσουμε να εντάξουμε σε αυτή τη δική μας γνωμοδότηση. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία έχω προτάσεις για βελτίωση της έκθεσης. Την έκθεση τη βρίσκω καλή και ο εισηγητής έχει μία προσέγγιση που μπορούμε να υποστηρίξουμε όλοι νομίζω. Έχω όμως κάποιες προτάσεις για το πώς να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι είναι θετικό το ότι υπάρχουν οι δημοσιονομικές προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, περισσότερο μακροπρόθεσμο από ό,τι σε πολλά κράτη-μέλη. Ένα από τα προβλήματα με τη χρήση πόρων σε πολλές χώρες είναι ότι ακολουθούν πολύ βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό. και πολύ συχνά έχουν ε, καινούρια οικονομική πολιτική κάθε χρόνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μακροπρόθεσμη προοπτική και γι' αυτό μας χρειάζονται κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τις βασικές δομές μακροπρόθεσμα και πρέπει να το κάνουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν, έχουμε, αν λάβουμε κακές αποφάσεις ε, με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο σοβαρές πρέπει να τονίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σίγουρα δεν πρέπει να υποστηρίζει μέτρα στα κράτη-μέλη τα οποία θα είναι επιζήμια για το περιβάλλον και για το κλίμα. Και δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πολλά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξουν προγράμματα που αντιβαίνουν στους στόχους για το περιβάλλον και για το κλίμα. Αυτή είναι λοιπόν η βασική μας προσέγγιση σε αυτήν την έκθεση, ότι θέλουμε να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά. Ακόμη σκεφτόμαστε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε ως θετικό μέσο για να επιτύχουμε αλλαγές στα κράτη-μέλη. Η κοινή γεωργική πολιτική, παραδείγματος χάρη, είναι ένας τομέας όπου νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πολλές δυνατότητες. Και πρέπει στις προτάσεις μας, μέσα στη γνωμοδότηση αυτή, ε, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη για να διατίθεται η χρηματοδότηση για το περιβάλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το τι πρέπει να γίνει δηλαδή στην πράξη. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν όρια στο πόσο λεπτομερής μπορεί να είναι αυτή η έκθεση. Όταν μιλάμε όμως για την γεωργική πολιτική πρέπει να λάβουμε υπόψη το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας και γι' αυτό καλό θα ήταν να δώσουμε πρακτικές προτάσεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε στην πράξη συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι σε άλλες επιτροπές αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα σε σχέση με την έκθεση αυτή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πολλοί περιβαλλοντικοί δείκτες και πρέπει να τονίσουμε ότι στην Επιτροπή μας πιστεύουμε ότι στην όλη συζήτηση ε, που αποκαλούμε πέρα από το ΑΕΠ λαμβάνουμε υπόψη και τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που έχουν σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική. Αυτές είναι προς το παρόν οι παρατηρήσεις μου. Θα σας δώσω και γραπτός βέβαια πολλά στοιχεία από αυτά που είπα. Πιστεύω ότι είναι μια καλή προσέγγιση και η έκθεση θα είναι εξαιρετική η έκθεση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φεραίρο, Ζεο Α, όχι, λάθος κάνω λέει πρόεδρος. Φερνάντες, συγγνώμη, συγγνώμη. Φερνάντες, έκανα εγώ λάθος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τους εισηγητές για το έργο τους. Έχω κάποιες προτάσεις για την έκθεση. Οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα βασιστούν στους ε, στόχους της στρατηγικής μας για το 2020. Θα έπρεπε να αναφέρεται η στρατηγική αυτή του 2020 και να φαίνεται ότι υπάρχει ο σαφής στόχος μας που είναι το 20-20-20. 20% μείωση δηλαδή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, 20% επίσης αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 20% αύξηση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ανανεώσιμων μάλλον πηγών ενέργειας. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε, να είναι σαφές, να φαίνεται. Και επιπλέον αυτή η στρατηγική υποστηρίζει μια πρωτοβουλία που απαιτεί χρηματοδότηση. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει και αποτελεσματικότητα όσον αφορά τους πόρους με τους οποίους χρηματοδοτούμε τη στρατηγική αυτή. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε λέγοντας κατά πόσο συμφωνούμε ή όχι με την στρατηγική αυτή. Αυτό θέλω να πω εγώ σχετικά με την γνωμοδότηση. Και κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Και Παντού πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, αλλά στον τομέα του περιβάλλοντος ακόμα περισσότερο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι που πάνε τα χρήματα σε ποιο σχέδιο, σε ποιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται όσο γίνεται καλύτερα και να ξέρουμε κατά πόσο η χρήση τους γίνεται σωστά και αποδοτικά. Είναι σημαντικό λοιπόν με τις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές να γίνεται σαφής η χρήση των πόρων αυτών υπέρ της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Η κυρία Χάγκα έχει τώρα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Πρέπει να πω, καταρχήν δεν έχω πολλά να πω για την έκθεση του κ. Γκεμπράντη. Όπως είπε και ο Ζωζέ Μανουέλ μόλις τώρα, μας ενδιαφέρει μια ενδυνάμωση, μια, ολοκληρωτική, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. στο Κοινοβούλιο βασιζόμαστε στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Θέλουμε έξυπνη, βιώσιμη και πολυσυλλεκτική ανάπτυξη που δεν αποκλεί κανέναν. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση στο δικό μας τομέα, στον τομέα του περιβάλλοντος και να έχουμε ένα στόχο σε μια πολιτική. Μπορεί ένα στόχος από τους τρεις να πρέπει να προωθηθεί περισσότερο, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τους άλλους δύο. Και αυτό πρέπει να το φροντίσουμε λίγο στην έκθεση. Και σαφώς η γεωργική πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και η πολιτική συνοχής. Και θέλω ήδη από τώρα να καλέσω όλους τους συναδέλφους στις 13 Ιανουαρίου να έρθετε στην Επιτροπή, στην Επιτροπή ΣΟΥΡ, όπου θα αρχίσουμε να ασχολούμεθα με τα τομεακά θέματα. Και στις 13 Ιανουαρίου ξεκινάμε με την γεωργική πολιτική. Θα ήταν εξαιρετικό το να μην έχουμε μόνο τους υπευθύνους της γεωργικής πολιτικής, αλλά να ακούσουμε και την, ε, τους εκπροσώπους της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής για να εκφράσουν όλοι αυτά τα οποία τους απασχολούν και αυτά τα οποία επιθυμούν και να πούν ότι στο αβ σημείο θέλουμε να βάλουμε κάτι ή να αλλάξουμε κάτι. Ήδη έχουμε κάποια εικόνα για το πώς θα θέλαμε να έχουν τα πράγματα. Άρα αυτά μπορούμε να τα πούμε στις 13. Κάτι το οποίο κάπως λείπει είναι τι κάνουμε εμείς και εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, τι κάνουμε στη βοήθεια που δίνουμε για φυσικές καταστροφές. Αυτό θα το αφήσουμε εντελώ απ' έξω, δεν θέλουμε να το αναφέρουμε καθόλου. Ή μήπως στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θέλουμε να το θίξουμε και αυτό. Ή έχουμε κατά νου ένα εντελώς διαφορετικό εργαλείο. Είναι μια σκέψη που πρέπει να μας απασχολήσει. Έχουμε χρόνο βέβαια. Όσον αφορά το έγγραφο εργασίας, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι κάπως υπερβολική διατύπωση strongest tool, το πιο ε, ισχυρό εργαλείο που έχουμε για το περιβάλλον. Η νομοθεσία μας είναι το πιο ισχυρό εργαλείο και ενδεχομένως και η συνεργασία πριν από τον προϋπολογισμό. Μέχρι τώρα στις τωρινές δημοσιονομικές προοπτικές ε, δεν μας είχαν δώσει τόσο πολλά χρήματα. Γι' αυτό θα προτιμούσα την ολοκληρωμένη προσέγγιση στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και μια τελευταία παρατήρηση. Όταν μιλάμε για έξυπνη ανάπτυξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φροντίσουμε όχι μόνο τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, αλλά και την παιδεία, ε, εκπαίδευση και κατάρτιση. Στο σημείο 7 κάπως αναφέρεται, κάπως θίγεται αυτό το θέμα. Γιατί λέει ο Γκέμπεν για εκεί επαρκεί πόρους για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Αλλά νομίζω ότι κάτι παραπάνω πρέπει να πούμε εκεί. οι καλύτεροι στόχοι δεν θα μας ωφελήσουν αν δεν έχουμε μέσα στα κράτη-μέλη επαρκείς ανθρώπους ε, που θα σκέπτονται έχοντας κατά νου την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να στραφούν ε, από τη σκέψη τους μόνο υπέρ του μέγιστου κόστους στη σκέψη τους ε, υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε, να επανακαταρτήσουμε ε, όλους, γιατί όταν ε, βάζουμε στην κατάρτιση, παραδείγματος χάρη ένα πρόγραμμα για τους ε, μηχανικούς, θα πρέπει να, να συμπεριλαμβάνεται στην κατάρτισή τους κάτι που θα τους κάνει να σκέπτονται με τρόπο βιώσιμο στο μέλλον. Κάτι παραπάνω χρειάζεται. Ελπίζω, ε, θα έλεγα, να γεμίσουμε τη σελίδα τουλάχιστον. Αυτά που έχουμε να συμπεριλαμβάνουν λίγο περισσότερα ε, στοιχεία. Αυτοί οι στόχοι πάντως που υπάρχουν εδώ, νομίζω ότι και στην Επιτροπή ΣΟΥΡ μπορεί να γίνουν αποδεκτοί. Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Γκέρμπεν Γιάνν Γκερμπράντι και τη Γιούτα Χάουγκ, που είναι η πιο σημαντική μορφή σε αυτή τη συζήτηση που πάντοτε συνεργάζεται με την Επιτροπή μας με επικοδομητικό τρόπο. Το 2005 αποφασίστηκαν οι τελευταίες δημοσιονομικές προοπτικές. Το 2007, όπως είπε ο συνάδελφος ε, Φερνάντες, ε, αποφασίσαμε τη στρατηγική 2020-2020. Και τώρα θα πρέπει ε, να προσαρμόσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές σε αυτή τη στρατηγική. Και πρέπει να πω ότι ε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, είπαμε την περασμένη εβδομάδα που αποφασίσαμε το 30%. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, ε, το ΕΛΚ μπορεί να πιστεύει ότι δεν είναι ε, όριμος ακόμη ο χρόνος, αλλά για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές σίγουρα θα πρέπει να έχει οριμάσει η περίοδος για να φτάσουμε στο 30% και είναι κάτι που πρέπει να το εντάξουμε στις προσπάθειές μας για το κλίμα. Ε, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Για να φτάσουμε το 30% χρειάζεται να έχουμε και επαρκείς οικονομικούς πόρους και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί στα κράτη-μέλη ε, ένας τρόπος και εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο υποστήριξης προ τα κράτη-μέλη ε, και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη αρκετά φιλόδοξου στόχου, να τα βοηθήσουμε να κάνουν πιο φιλόδοξου τους στόχους τους για το κλίμα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε όχι μόνο τη βραχυπρόθεσμη συζήτηση, τώρα μπορεί να δυσκολευόμαστε στα θέματα αλλαγή του κλίματος και να βλέπουμε ότι δεν επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, γιατί αν θέλουμε να το κάνουμε κάτι και στους στόχους του ΕΛΚ υπάρχει αυτό, πρέπει στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να εκφράζεται κιόλα. Ευχαριστώ, Πέτερ. Γιάν, ένα σύντομο συμπέρασμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ναι, θα είμαι σύντομο. Συμφωνώ πάρα πολύ με όλα τα σχόλια περίπου των συναδέλφων. Ενισχύουν τα όσα και εγώ έχω συμπεριλάβει. Σας είπα και πριν ότι δεν είχα αρκετό χώρο να τα βάλω όλα. 20-20-20. Ναι, πρέπει να αναφέρεται ρητά. Όπως επίσης και Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Η διαφάνεια του κύριου Φερνάντες, ναι, πάρα πολύ σωστό, Ξέρετε το σημείο. Να το συμπεριλάβουμε. Τι άλλο. Το θέμα της ε, παράτασης αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. πρέπει το μήνυμα της γνωμοδότησης να παραμείνει ισχυρό. Σας είπα ότι ήθελα από τους συναδέλφους να με βοηθήσουν και να επεκτείνω κάπως το κείμενο, αλλά και να το καταστήσω πιο ισχυρό και νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, δουλειά σας. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 14 Δεκεμβρίου. 26 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση και τον Μάρτιο τον Απρίλιο του 2011 θα πάει στην Ολομέλεια προς ψήφιση η έκθεση. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Έληξε συνεδρίαση.